then I, will indicate it. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα καλωσορίσω στη σημερινή μας συνεδρίαση της επιτροπή Έλεγχου του Βλέπετε πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή μας, γιατί σήμερα έχουμε πάρει αυτή τη μεγάλη αίθουσα ίσως ε, λόγω της μεγαλύτερης προσοχής που περιστρέφεται γύρω από το έργο μας, εν πάση περιπτώσει το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της και επομένως εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή όλα αυτά τα θέματα. Τώρα να περάσουμε τα τυπικά θέματα. Έχετε την ημέρησια διάταξη. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Γενικός ε, Διευθυντής της Όλαφ με μια επιστολή προς την Επιτροπή μας ζήτησε να μπορέσει να μας πληροφορήσει για την κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με, την, ε, με τα θέματα της Επιτροπής Παρακολούθησης και επίσης έχουμε τα ζητήματα της ε, διαθεσμικής ε, συνεργασίας των μεγάλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά και είπαμε στον κύριο ε, επικεφαλής της ΟΛΑΦ ότι θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή την παρουσίαση και να ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις των βουλευτών της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής μας. Σα το λέω αυτό γιατί αυτό, αυτή η αίτησή του έγινε μετά από την σύνταξη και εκτύπωση της ημερησίας διάταξης. Υπάρχουν τώρα ερωτήματα για την ημερησία διάταξη, αντιρρήσει κτλ. Ούτως έχει αποφασιστεί. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι είναι ε, δημόσια συνεδρίασή μας και μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο, στο τρίτο σημείο, στην έγκριση των πρακτικών. Πρόκειται για τα πρακτικά της 6ης Νοεμβρίου 2012. Έχετε παρατηρήσει σχετικά. Εάν όχι, τότε θεωρεί ότι έχει εγκριθεί. Έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της 6ης Νοεμβρίου. Περνάμε στο σημείο 4. Απαλλαγή 2011, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα 3, Επίτροπη. Θα ήθελα σχετικά να χαιρετήσω την παρουσία του Επιτρόπου για την Γεωργία, του κυρίου Τσόλος. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι σήμερα του Αγίου Νικολάου. Ίσως αυτό έχει και κάποιο συμβολικό χαρακτήρα, γιατί φυσικά η ημέρα του Αγίου Νικολάου είναι και το αντίστοιχο για τα ελληνικά δεδομένα της ε, ημέρας του Αγίου Βασίλη. Είναι ο, ο Άγιος Βασίλης των Γερμανών, ο Άγιος Νικόλαος και θα μας φέρετε, ελπίζω, δώρα τα οποία μπορεί να είναι υπό τη μορφή τροφίμων, γιατί για πολλά μέρη του κόσμου τα τρόφιμα δεν είναι πια κάτι το δεδομένο. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε μια επιτυχή <clears throat> πολιτική για τα αγροτικά θέματα που θα εξασφαλίσει μια σωστή διατροφή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε και μια εξαγωγική δύναμη σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα. Σήμερα πρόκειται για τεχνικές ρυθμίσεις για τα θέματα της γεωργίας και επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου και θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Αγκουστίν Κούμπικ και τον κύριο Ράσα Μπουτμπιγκέρτη να χαιρετήσω στο Ευρωπαϊκό, στην ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας και θα τους δώσω στη συνέχεια το λόγο. Ξεκινώ λοιπόν με τον εισηγητή κύριο Γκάιερ και μετά θα δώσω το λόγο σε εκπροσώπους του Ελεκτρού Συνεδρίου. Κύριε Γκάιερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και από μένα καλημέρα σε όλους. Εγώ θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Τσόλος για την παρουσία του και για την διαθεσιμότητά του να ανταλλάξει απόψεις μαζί μα. Και επίση χαιρετίζω τα διακεκριμένα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε ορισμένα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την απαλλαγή από τον προϋπολογισμό του 2011. Καταρχήν τα θέματα του προϋπολογισμού στην ε, αγροτική πολιτική που αν πάρουμε και, τις, και τους δύο πυλώνες της ε, Γεωργίας είναι ακόμα η μεγαλύτερη παρτίδα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη σωστή εξέλιξη του αγροτικού τομέα πέραν του τομέα της έρευνας ο τομέας της ε, γεωργίας είναι ένας τομέας όπου τα επίπεδα σφαλμάτων στον προϋπολογισμό του 2011 έχουν ανέλθει, έχουν αυξηθεί τα σφάλματα αντί να μειωθούν. Έχουμε ένα ποσοστό σφαλμάτων στην αγροτική ανάπτυξη που έχει φτάσει σε ένα ανισχυτικό επίπεδο 7,7% σφαλμάτων. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό μας γεννά πολλές ανησυχίες. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για τα θέματα της ε, περιφερειακής πολιτικής, είναι σημαντική η ανάλυση στην οποία έχει προβεί το ελεκτικό συνέδριο που τονίζει ότι πολλά προβλήματα έρχονται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς των κρατών μελών και η άνοδος των σφαλμάτων στον τομέα αυτό της γεωργίας δείχνουν ότι υπάρχει και εδώ ένα πρόβλημα που έχουμε δει σε άλλους τομείς και αυτό μας ενοχλεί ιδιαίτερα γιατί στις διαπραγματεύσεις ε, για, την, ε, για τις δημοσιονομικές προοπτικές στην επόμενη επταετία βλέπουμε από την πλευρά του Συμβούλιου μια θέληση να περισταλούν ε, τα κονδύλια στον γεωργικό τομέα με το πρόσχημα ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με μια καλύτερη διαχείριση των better spending όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Και η δική μου απάντηση στα θέματα αυτά είναι ότι τα στοιχεία στον αγροτικό τομέα δείχνουν ότι όποιος θέλει καλύτερη διαχείριση, better spending, θα πρέπει να ξεκινήσει από το σπίτι του, από την, το δικό του χώρο με καλύτερο έλεγχο στα αγροτικά κονδύλια. Θα θέλαμε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε με τον κύριο Επίτροπο για το πώς τα θέματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν και να τακτοποιηθούν το ταχύτερο. Εμείς θα πρέπει μέχρι τον Απρίλιο, κανονικά μέχρι τον Μάιο, αλλά αυτή τη φορά μέχρι τον ε, Μάιο, μέχρι τον Απρίλιο αυτή τη φορά προβλέπεται. Η απαλλαγή πρέπει βάσει των συνδικών να δοθεί μέχρι τις 15 Μαΐου και επειδή δεν έχουμε την αίθουσα της Ολομέλειας Βρυξέλλες πια θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη ε, διαδικασία απαλλαγή στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Αυτό μας δίνει κάποια πίεση, έχουμε μια πίεση χρόνου και επομένως εδώ χρειάζεται να ληφθούν ορισμένε αποφάσεις. Θα πρέπει να δώσουμε την απαλλαγή στην Κομισιόν για την εκτέλεση του προπολογισμού του 2011. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι η Κομισιόν πράττει όλα τα απαραίτητα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί σε αυτόν τον ζωτικό τομέα. Και γι' αυτό είναι μια μεγάλη χαρά για μας που μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσόλος. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω εδώ και θα περιμένω να ακούσω τις απόψεις του ελεκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Στρέφομαι λοιπόν προς το ελεκτικό συνέδριο. Δεν, δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει, ο κύριος Κούμπικ ή η κυρία Μπουτμπεργίτα. Κύριε Κούμπικ καταρχήν. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για μας να σας παρουσιάσουμε την προσπάθεια την οποία ολοκλήρωσε το ελεγκτικό συνέδριο στην άμεση στήριξη στη Γεωργία στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης για το 2011. Καλύπτουμε τις δαπάνες από το Ταμείο Εγγυήσεων που έφτανε περίπου στα 44 δις ευρώ το 2011 και αντιπροσωπεύει άνω του 1 τρίτου του ε, προϋπολογισμού της κοινότητας φέτος για πρώτη φορά Κάναμε δύο διαφορετικές ε, αξιολογήσεις, μία για το HEF και ε, μία δεύτερη για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό το κάναμε για να ανταποκριθούμε στο αίτημα των αρχών απαλλαγής έτσι ώστε να δούνε καλύτερα το περιεχόμενο των δύο πολιτικών. Να έρθω λοιπόν στα βασικά συμπεράσματα της έρευνές μας. Τα βασικά λάθη των πληρωμών για το 2011 φτάνει περίπου στο 2,9%. Το ποσοστό αυτό βασίζεται στην αξιολόγηση και στον έλεγχο 208 πληρωμών, κάποιων δειγμάτων δηλαδή από το σύνολο των πληρωμών. Βρήκαμε να υπάρχει πρόοδος στην νομιμότητα και στον τακτικό χαρακτήρα των πληρωμών και η κατάσταση πάνω κάτω όμως είναι στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο χρόνο σύμφωνα με το ε, σύστημα ελέγχου Άγιαξ το οποίο ισχύει για έξι αρχές πληρωμών. Νομίζω ότι η διαδικασία εμπολής διασφαλίζει τις, ανα... απαιτήσει οι οποίες υπάρχουν. Ας έρθω όμως συγκεκριμένα τώρα στα συγκεκριμένα ε, συμπεράσματα. Σχετικά με το ποσοστό λάθος. Τι λάθη καταρχάς εμείς βρήκαμε. Νομίζω ότι δεν εκπλήσεται κανείς όταν δει ότι η πλειοψηφία των λαθών είναι επιπλέον δηλώσεις ε, ε, περιοχών. Ένα μεγάλο ποσοστό του ταμείου αυτού είναι άμεσες πληρωμές προς τους ε, γεωργούς. Είναι 5% οι δηλώσεις οι οποίες έχουν επιπλέον επιφάνειες. το σύστημα εντοπισμού γεών το οποίο χρησιμοποιήθηκε μας βοήθησε να μειώσουμε τα περιθώρια λάθος. Τώρα πώς συγκρίνεται αυτό με το 2010. Πέρυσι είχαμε στοιχεία λάθος για το σύνολο της γεωργίας και για το ε, HF αλλά και για το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου. Το ποσοστό αυτό πέρυσι ήταν 2,3%. Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε το 2010 και το 2011, τα αποτελέσματά τους δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τον συνδυασμένο δείκτη λάθους και για τις δύο πλευρές αυτές που φτάνει το 4%. 0,2% του συγκεκριμένου ποσοστού λάθους δημιουργείται από κάποιες αλλαγές απλά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε σχετικά με τις παραβιάσεις των τομέα in a minute. So in real terms... Της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η αύξηση του ποσοστού των λαθών από το 2010 μέχρι το 2011 είναι 1,5%. Από 2,3% περάσαμε ουσιαστικά στο 3,8%. Αυτή η αύξηση του 1,5% είναι σημαντική αύξηση. Η αύξηση αυτή όμως θα πρέπει να γίνει αντικείμενο ερμηνείας με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το μεγαλύτερο ποσοστό εξήγησης θα έλεγα είναι ανάμεσα στις ανώτατες και στις πολύ χαμηλές ε, ε, εννοώ ποσότητες και δηλώσεις. Σαν ελεγκτής θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να περιμένουμε κάποια χρόνια ακόμα για να δούμε αν το σημερινό ποσοστό είναι μια φυσιολογική και αναμενόμενη στατιστική διακύμανση ή πράγματι αποδεικνύει ότι υπάρχει μια συνολική χειροτέρευση αν θέλετε του συστήματος πληρωμών. Ε, τα στοιχεία που θα έχουμε για το 12 του χρόνου θα μας δώσουν περισσότερες δυνατότητες να ερμηνεύσουμε το θέμα. Τώρα για την πολλαπλή συμμόρφωση πώς εμείς τροποποιήσαμε τον τρόπο που λειτουργούσαμε μέχρι τώρα. Όπως είπα το 2011 για πρώτη φορά το ε, ελεγκτικό συνέδριο ε, συμπεριέλαβε τις παραβιάσεις της πολλαπλής ε, συμμόρφωσης. Τέτοιου είδους παραβιάσεις επηρεάζουν τις συνθήκες καταβολής των πληρωμών. Όλοι οι εποφελούμενοι από την κοινοτική βοήθεια θα πρέπει να σέβονται τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης. Εάν οι γεωργοί αποτύχουν στην προσπάθεια σεβασμού αυτών των απαιτήσεων, τότε μειώνεται η βοήθεια την οποία λαμβάνουν. Να υπογραμμίσω ότι για λόγους τεχνικούς και για λόγους εφικτότητας, οι ελεγκτικές διαδικασίες του συνεδρίου δεν καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις ε, της πολλαπλής συμμόρφωσης και γι' αυτό περιοριστήκαμε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Όπως είπα, οι επιπτώσει του ποσοστού λάθους για αυτές τις επιλεγμένες απαιτήσει στον τομέα της πολλαπλής συμμόρφωσης ανέρχονται στο 0,2%. Όμως, λόγω ακριβώς των περιορισμών ε, που έχουν τεθεί στην εμβέλεια των ελέγχων για την πολλαπλή συμμόρφωση, θα πρέπει το ποσοστό αυτό να το χρησιμοποιήσουμε με πολύ επιφυλακτικότητα και να μην θεωρήσουμε ότι είναι μια γενικότερη κρίση του συστήματος πληρωμών προς τους γεωργούς. Τώρα για την αξιολόγηση των συστημάτων. Εμείς αξιολογήσαμε τα συστήματα αυτά και σχετικά με το σύστημα Ajax Είδαμε ότι το σύστημα πληρωμών στις υπηρεσίες τις εξωτερικές τις οποίες επισκεφθήκαμε επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται και από τις διάφορες μορφές δεδομένων οι οποίες ελέγχονται. Από τις επιφάνειες όπως επίσης και από λανθασμένες καταθέσεις στοιχείων. Ε, κάποιες, κάποια συστηματικά λάθη στη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου έχουν διαπιστωθεί και ήδη ε, κάποια προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια δεν διορθώθηκαν και συνεχίζουν να οδηγούν σε μη κανονικές πληρωμές. Τέτοιες αδυναμίες εντοπίζονται σαν παράδειγμα στην ταξινόμηση της χρήσης των γεών ή στις επιπλέον ε, δηλώσεις στοιχείων στο σύστημα εντοπισμού ε, των γεωργικών επιφανειών και τη λανθασμένη ε, προφανώς εφαρμογή ορισμένων ενιών και ορισμών μάλλον. Έχουμε λοιπόν προχωρήσει ε, στον εντοπισμό λανθασμένων υπολογισμών γεωργικών γεών σε τρία χώρες μέλη οι μετρήσεις μας διαφοροποιούνται από τα αποτελέσματα τα οποία είχαν καταθέσει οι υπηρεσίες πληρωμών, οι αρχές πληρωμών. Ταυτόχρονα εμείς εξετάσαμε ε, και τις... Ε, και το σύστημα το οποίο οδηγεί στην κατάθεση των δηλώσεων αξιοπιστίας και είδαμε ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Λοιπόν αυτά είναι γενικότερα τα προβλήματα, ίσως να σταθώ τώρα σε κάποιες συστάσεις. Καταρχάς, αναγνωρίζουμε ότι ελήφθησαν ορισμένες δράσεις διορθωτικές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέτοντας ε, και κάποια επιπλέον ποιοτικά στοιχεία ελέγχου στο σύστημα εντοπισμού αγροτικών γεών, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό του ελέγχου των συστήματος πληρωμών. Παρ' όλα αυτά, στα πλαίσια των ευρημάτων, εμείς συστήνουμε σαν συνέδριο τα εξής. Η σωστή αξιολόγηση της επιλεξιμότητας μονίμων ε, χορτολιβαδικών εκτάσεων θα πρέπει να διασφαλιστεί οι αρχές πληρωμών θα πρέπει να διορθώσουν τα διοικητικά προβλήματα και τα ελεγκτικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν. Η ποιότητα των επιτόπου ελέγχων θα πρέπει να βελτιωθεί και τέλος, ο σχεδιασμός και η ποιότητα των προσπαθειών οι οποίες επιτελούνται από τα λεγόμενα εγκεκριμένα εξωτερικά σώματα θα πρέπει να μας επιτρέπουν να οδηγηθούμε στη σωστή αξιολόγηση των συστημάτων πληρωμών από τις εξωτερικές αρχές. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Thank you very much, Mr. Kubik. Ευχαριστούμε κύριε Κούμπικ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μπουτμπεγκέιτη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, με χαρά θα σα παρουσιάσω το κεφάλαιο 4 τη ετήσια έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου το 2011, το οποίο αφορά δηλαδή ανάπτυξη υπέδρου περιβάλλον, υγεία, λία. Όπω ε, ο συνάδελφό μου κύριο Κούμπικ μόλι προανέφερε, πρόκειται για πρώτη φορά όπου αφιερώνεται εσείς ε, στο μισό ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι 13,9 δις ευρώ, δηλαδή 10,7% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, των οποίων ε, η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι το 12,4 δις ευρώ. Οι δαπάνε στον τομέα αυτό βασίζονται σε συγχρηματοδότηση και καλύπτουν μέτρα σχετιζόμενα με τις περιοχές και όχι τόσο σχετιζόμενα με τις ε, περιοχές. Τα πρώτα που σχετίζονται δηλαδή με τις περιοχές είναι γεωργοπεριβαλλοντικά ε, συστήματα, σχήματα και αυτά που δεν σχετίζονται είναι επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό. Πού καταλήγουμε ως συνέδριο είναι ότι πληρωμές για το 2011 για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για το περιβάλλον, για την αλληλεία, για την υγεία επηρεάστηκαν αποσιαστικά σφάλματα τα συστήματα ελέγχου και επαλήθευσης ήταν λοιπόν εν μέρη αποτελεσματικά μόνο. Γιατί καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό για τις ε, συναλλαγές και για τα συστήματα. Σε ό,τι αφορά τις ε, δοκιμές για τις συναλλαγές, για τις πράξεις, ε, πήραμε ως δείγμα 178 ενδιάμεσες και τελικές απληρωμές, από τις οποίες 160 φορούσαν τις πληρώμες αυτές για την αγροτική ανάπτυξη. Στο ποσοστό των σφαλμάτων βλέπουμε πολύ ψηλότερα επίπεδα για την αγροτική ανάπτυξη σχέση με τους άλλους τρεις τομείς και κυρίως ε, φτάσαμε σε αυτό το ποσοστό του 7,7% το οποίο παραπέμπει και στη δήλωσή μας περσινής χρονιά ότι στον τομέα αυτό δηλαδή της ανάπτυξης πέτρου έχουμε σημαντικά περιθώρια ασφάλματος και κυρίως πρόκειτο για την επιλεξιμότητα μέτρων μη σχετιζόμενων με τις περιοχές εν μέρη λόγω των σχετικά πολύπλοκων συνήθως κανόνων και των κριτήριων επιλεξιμότητας για τα μέτρα αυτά. Τα σφάλματα αυτά οφείλονται λοιπόν στο γεγονός ότι το ίδιο το project, το ίδιο το έργο ή μέρος του ή ακόμη και ο δικαιούχος δεν ήταν επιλέξιμος δυνάμει ε, των, των κανόνων που ισχύουν για τα μέτρα αυτά. Κάποιε φορέ μάλιστα δικαιούχοι ήταν δημόσιοι οργανισμοί ή ήταν και οι ίδιοι ω οργανισμό πληρωμή. Όπω συνέβη στην περίπτωση όπου οι διαδικασίε ε, δημόσιων διαγωνισμών, δημόσιων συμβάσεων εφαρμόζονται. Δηλαδή βλέπουμε να μην ακολουθούνται, να μην τηρούνται πάντοτε οι διαδικασίε. Για παράδειγμα, για την ε, απόφαση περί ανάθεση συμβάσεων με διαδικασίε άλλε, όχι ανοιχτού διαγωνισμού. Βλέπουμε εκεί να μην δικαιολογείται αυτή η προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία σε πολλέ περιπτώσει. Τώρα, για μέτρα σχετιζόμενα με τις περιοχές, ε, τα περισσότερα αφορούσαν ε, γεωργοπεριβαλλοντικά σχήματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι αγρότε δεν είχαν σεβαστεί τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσει, τι οποίε είχαν αναλάβει και που αποτελούσαν και συχνά την προϋπόθεση για την πληρωμή Επίσης είδαμε σφάλματα πολλαπλής συμμόρφωση στο 66% σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή των υποχρεώσεων για την ε, πολλαπλή συμμόρφωση. Για πρώτη φορά ως ε, συνέδριο ποσοτικοποιήσαμε τα σφάλματα. 0,2 είναι το ποσοστό σε σχέση με το 7,7 συνολικά, δηλαδή ποσοστό σφάλματος για το κεφάλαιο 4 και αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση αυτό το 0,2. Είδαμε δηλαδή προβλήματα, παραδείγματο χάρη για την καταγραφή, την καταχώρηση των ζώων. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τι δοκιμέ ε, στι πληρωμέ ε, για το περιβάλλον, την αλία και ε, την δεν βλέπουμε σημαντικέ, ε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, διότι είχαμε μόνο 18 ελέγχους. Ό,τι αφορά τώρα τα εποπτικά ελεγκτικά συστήματα, Ελέγξαμε σε έξι χώρες μέλη τα συστήματα σε ό,τι αφορά την εκαθάριση λογαριασμών, ε, τη διαχείριση, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΤΑ. ελέγξαμε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα ανάπτυξης υπαίθρου, ε, κάναμε ελέγχους σε, μία ε, οργάνωση, σε έναν οργανισμό πληρωμών στις έξι χώρες ο ένας οργανισμός δεν ήταν αποτελεσματικός, οι τέσσερις ήταν εν μέρει αποτελεσματικοί και ο ένας ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή ε, εξασφαλιζόταν με αυτό η κανονικότητα των πληρωμών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα διοικητικά ελεγκτικά συστήματα, τα μελετήσαμε για να δούμε αν υπάρχουν σωστέ σωστές διαδικασίες καταβολής των πληρωμών. Είχαμε επιτόπιους ελέγχου και εφαρμόσαμε και συστήματα για να δούμε αν υπάρχει υλοποίηση και έλεγχος της πολλαπλής συμμόρφωση Τώρα, σε ό,τι αφορά το γάμα δέλτα άκρη για την ε, καθάριση των οργανισμών, το σύστημα τη εν περιλαμβάνει ελέγχου που διεξάγονται από ανεξάρτητου φορεί πιστοποίηση. Ε, το συνέδριο αναθεώρησε 32 ε, φορείς πιστοποίησης ως δείγμα και βρήκε ότι οι παρατηρήσεις τις οποίες είχαμε επισημάνει σε προηγούμενους ελέγχους συγκεκριμένα που είχε διεξαγάγει η Κομισιόν βλέπουμε διαπιστώνονται η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη δεν ε, προέβη στους σωστούς έλεγχους, δεν επαλήθευσε αυτά τα, αυτές τις παρατηρήσεις, ούτε τις έλαβε υπόψη τη σε ό,τι αφορά τη σχέσεις πεπραγμένων. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανάλυση, δεν υπάρχει εξήγηση του γιατί οι πολυματικά ποσοστά σφαλμάτων για την ε, αγροτική ανάπτυξη αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο, όπως λέει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το ποσοστό σφαλμάτων ήταν πολύ χαμηλότερο σε σχέση με του ε, συνεδρίου, διότι βασιζόταν σε στοιχεία τα οποία είχαν δώσει τα κράτη-μέλη για το 2010. και όπως ε, λέμε ε, δεν ε, ανοιχνεύτηκαν ούτε αναφέρθηκαν όλες οι μη επιλέξιμες δαπάνες από τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν αδυναμίες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των οργανισμών καταβολής πληρωμών. Για τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ τώρα οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπήρχε πλήρης τεκμήρωση για όλους τους βασικούς ελέγχους, ούτε επαρκής επιτήρηση και επαλήθευση, ιδίω ό,τι αφορά το τομέα των διεθνών ε, αλληλευτικών συμφωνιών. Για να βοηθήσουμε λοιπόν να διορθωθούν αυτά τα συστήματα, έχουμε ένα ε, σύστημα, το... μάλλον έχουμε τις εξή συστάσεις. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη απλούστευση των κανόνων. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου με πιο αυστηρό τρόπο. Επίσης, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι φυστάμενοι κανόνε ε, εφαρμόζονται καλύτερα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά τι γεωργοπεριβαλλοντικέ δεσμεύσεις και την επιλεξιμότητα για μέτρα επενδυτικά. Επίση, το συνέδριο συνιστά η Κομισιόν να αναλύσει του λόγου για αυτό το πολύ σημαντικό ποσοστό σφαλμάτων και να εξασφαλίσει ότι η δέλτα άγκρη και οι φορείς πιστοποίησης θα λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα προηγούμενων ελέγχων που έχει διενεργήσει η Κομισιόν και το συνέδριο για την εκπόνηση των στρατηγικών ελέγχων. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας και με τα θα απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπεντουαγκίτα για την εκθεσή σας. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω τον ε, Επίτροπο ή αν θέλει ο εισηγητής να παρέμβει προηγουμένως. Όχι, ο Επίτροπος ε, Τσόλος έχετε ακούσει την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την Επιτροπή μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιες απαντήσεις ιδίως για την διαφαινόμενη αύξηση των σφαλμάτων στην αγροτική ανάπτυξη. Βέβαια είναι μικρή αυτή η αύξηση από τη μια μεριά, αλλά υπάρχουν πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και ίσως θα μπορούσατε να μας απαντήσετε για τα θέματα αυτά. Καλώς ήλθατε και πάλι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Συγητή επίσης, ε, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, έντιμα μέλη της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού Χαίρομαι που μπορώ να λάβω το λόγο μετά από την παρουσίαση της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου για να διευκρινίσω ορισμένα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να το πράξω αυτό διότι προετοιμάσουμε και μία μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής που είναι μια ευκαιρία να προχωρήσουμε για τους πολιτικούς μας στόχους στον τομέα της αγροτικής πολιτικής αλλά για να εξασφαλίσουμε και την καλύτερη διαχείριση των πόρων στην αγροτική αυτή πολιτική. Επομένως θα πρέπει όλοι να αντλήσουμε διδάγματα από το έργο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Για πρώτη φορά το ελεκτικό συνέδριο, όπως ελέγχθη, έχει αφιερώσει δύο κεφάλαια στις δαπάνες της κοινή αγροτικής πολιτικής και έχει δώσει δύο διαφορετικά ποσοστά για τα σφάλματα. Ένα για τον πρώτο πυλώνα των εγγυήσεων και το δεύτερο για τον πυλώνα των ε, δομών της αγροτικής ανάπτυξης. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τα 80% περίπου των αγροτικών δαπανών όπως ανέφερε και ο κύριος Κουμπίκ. Για πρώτη φορά το ελεκτικό συνέδριο έλαβε υπόψη τις, ε, τα ασφάλματα που έχουν να κάνουν με την πολλαπλή συμμόρφωση. Είναι σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία για την συνεχή βελτίωση των συστημάτων στον αγροτικό τομέα και για μένα αποτελούν ένα σημαντικό μήνυμα γιατί οι πληρωμές στον αγροτικό τομέα είναι ένα σημαντικός πολιτικός μοχλός ανάπτυξης για την απασχόληση και την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι επίσης και ένα σημαντικός μοχλός και παράγοντας για την προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, έχω λάβει υπόψη όλα αυτά τα οποία ανέφερε το ελεκτικό συνέδριο. Είναι σαφές ότι οι προσπάθειες οι οποίες έχουν καταβληθεί για το LPAS, για τον εντοπισμό των αγροτικών αγροτεμαχίων, θα συνεχιστούν και ιδίως με τη συνεργασία των χωρών που εξακολουθούν να έχουν προβλήματα στον τομέα αυτό. Βλέπω επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριμένε περιπτώσεις όπου τα ασφάλματα ήταν χαμηλότερα από 2%. Και οι δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν που υπήρξαν υψηλά ποσοστά ασφαλμάτων δεν καταδεικνύουν να υπάρχουν συστημικά προβλήματα. Πιστεύω ότι και στι δύο περιπτώσει με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των αρμοδίων κρατών μελών θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση. Και έρχομαι τώρα στους δύο πυλώνες όπου δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το επίπεδο των σφαλμάτων. Δύο διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι χρήματα τα οποία έχουν απολεστεί για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ούτε περιπτώσεις απατών στις περισσότερες περιπτώσεις που είδαμε σφάλματα να υπάρχουν. Δεύτερον, βρισκόμαστε και σε ένα επίπεδο κορύφωση σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των αγροτικών προγραμμάτων και είναι πιο λογικό να υπάρχουν περισσότερα σφάλματα από ό,τι στην αρχή της περίοδου προγραμματισμού όταν απλώς υπάρχει η προετοιμασία των σχεδίων και όχι η εκτέλεσή τους. Αυτό φυσικά δεν εξηγεί το επίπεδο των σφαλμάτων. Γι' αυτό χωρίς να περιμένουμε εμείς το τελικό έγγραφο της, ε, του ελεκτικού συνεδρίου έχουμε θεσπίσει μια, ένα αποθεματικό για το 2012 σε σχέση με τα θέματα αυτά. Μαζί με τις αγροτικές υπηρεσίες των κρατών μελών έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες μου να εξετάσουν τους λόγους για αυτή την κατάσταση. Η ανάλυση που έγινε κατέδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος των σφαλμάτων έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχει λάβει χώρα η, ο προγραμματισμός σε επίπεδο κρατών μελών. Είδαμε πολλά στοιχεία μεταξύ των οποίων εγώ θα ήθελα να αναφέρω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, οι προποθέσει επιλεξιμότητας πολλές φορές χρησιμοποιούνται Ε, αντί για την δέσμευση των ε, δικαιούχων. Υπάρχει λοιπόν ένα σφάλμα το οποίο καταμετράται ε, Θεωρείται ότι αυτό είναι ένα ε, στοιχείο δέσμευση των δικαιούχων, ενώ τα κράτη-μέλη το καταγράφουν μονάχα στον τομέα τη επιλεξιμότητα. Αυτό οδηγεί σε σφάλματα 100%. Επίση, πολλέ φορέ ο εντοπισμό των δικαιούχων είναι δύσκολο γιατί τα κριτήρια δεν έχουν διατυπωθεί σαφώ. Αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερο κίνδυνο σφαλμάτων. Γιατί τα κράτη-μέλη δεσμεύονται υπέρ ενό δικαιούχου, χωρί όμω να διευκρινίσουν τι προποθέσει για τον δικαιούχο πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη λύση για τα θέματα αυτά. Ε, οι υπηρεσίε μου έχουν ζητήσει να τροποποιηθούν ορισμένα προγράμματα, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει στη διάρκεια τη εκτέλεση των προγραμμάτων. Έχουμε ε, προσπαθήσει επίση να εξασφαλίσουμε και του ελέγχου συμμόρφωση για την εκτέλεση των δαπανών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Όλα αυτά θα μπορέσουν να αποδώσουν καρπούς από τον επόμενο χρόνο. Η νέα διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και να περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα λαμβάνουν από την αρχή την ανάγκη ελεξιμότητα των προγραμμάτων αυτών ανάπτυξη. ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλέ δράσει επίση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση που είναι εν εξελίξη και θα συνεχίσουν με τη βοήθεια και των κρατών μελών. Το θέμα αυτό εξάλλου βρίσκεται στη μέση διάταξη του πρόσφατου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και πληροφόρησα τους υπουργούς των κατών μελών για τα προβλήματα αυτά, ζητώντας τους να συνειδητοποιήσουν αυτές τις δυσκολίες και να αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα μαζί με την Επιτροπή. Θα δημοσιεύσουμε επίσης κατευθυντήρες γραμμές με θετικά και αρνητικά παραδείγματα γιατί υπάρχουν κάτι κράτη-μέλη τα οποία ήταν υποδειγματικά, αλλά είχαν προβλήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μάθουμε όλοι από τις βέλτιστες εμπειρίες στον τομέα αυτό. Η Κομισιόν επίσης έχει παίξει το ρόλο της ελέγχοντας τον βαθμό ελεγξιμότητος των κανόνων για την αγροτική ανάπτυξη και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε χρειάζονται χρόνο για να μπορέσει να υπενικηθεί μια κάποια αδράνεια που υπάρχει και για να αποδώσουν καρπούς θα πρέπει να περιμένουμε και τη νέα περίοδο προγραμματισμού για να δούμε να υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα, ακόμα και αν από τώρα εμείς θα πρέπει να ξεκινήσουμε με άμεσες δράσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. Προφανώς δεν θα περιμένουμε την επόμενη περίοδο προγραμματισμού για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ υποστη... βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ώστε η μεταρρύθμιση στον τομέα της κοινή αγροτικής πολιτικής και το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο θα επιφέρουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με τις κατάλληλες απαντήσεις στα προβλήματα για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση στον τομέα αυτό και φυσικά παραμένω στη διάθεσή σας για να απαντήσω τυχόν ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους βουλευτές οι οποίοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Ο κύριος Γκάιερος, εισηγητής πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και τον Επίτροπο Τσόλος για τις παρατηρήσεις τους. Καταρχήν, θέλω να θέσω τα εξή ερωτήματα στον κύριο Επίτροπο. Και θα ήθελα να σας πω ότι εμείς θα παρακολουθήσουμε μέχρι φυσικά την ημέρα της απαλλαγής, την στιγμή της ψηφοφορίας, τις ενέργειες που θα αναλάβουν οι υπηρεσίες σας για να άρουν τα προβλήματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί και να ξεκινήσουν την απαραίτητη διαδικασία για να μην υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στα επερχόμενα έτη. Αυτό θυμίζει λιγάκι ε, το γεγονός ότι αντίστοιχα με άλλους τομείς πολιτικής όπως είναι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να δώσουμε και μεγάλη έμφαση στα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το τομέα. Υπάρχει φυσικά το θέμα των ε, σφαλμάτων, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να τα λάβουμε υπόψη και να, να δούμε οι αναλύσεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε τι οδηγούν υπομορφή συμπεράσματος. Έχουμε ξεκινήσει μια πρακτική στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης η οποία έχει οδηγήσει και σε μια ανάγκη αντιπαράθεσης κατά κάποιο τρόπο με τα κράτη-μέλη που έχουν το υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων τα οποία έχουν διαπιστωθεί και είναι σαφές ότι αυτά δεν μας ικανοποιούν σε επίπεδο απόδοσης. Και είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουμε από πιο κοντά τα θέματα αυτά. Είχαμε πρόσφατα τον Υπουργό Αγροτικών Θεμάτων της Εχικής Δημοκρατίας ενώπιόν μας και αναφερθήκαμε στα θέματα της κρατικής διαχείρισης των ε, αγροτικών ταμείων ανάπτυξης και είχαμε μια ανταλλαγή απόψε για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Αυτό όμως σημαίνει ότι εμείς θα μπορούμε να ξέρουμε πού βρίσκονται τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα προβλήματα στα προγράμματα και εγώ ακριβώς γι' αυτό σας έθεσα το ερώτημα σε ποια κρατημέλη εστιάζονται τα παραδείγματα αυτά που ανέφερε το ελεκτικό συνέδριο. Θέλουμε να ξέρουμε που έχουν γίνει αυτά τα προβλήματα σε πιο κράτος μέλος και επίσης θα ήθελα να ξέρω αν μπορείτε για όλα αυτά τα θέματα που ανέφερε το ελεκτικό συνέδριο να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για να ξέρουμε ποια κρατημέλη θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πιο προσεκτικά και ενδεχομένω για να αποστείλουμε αποστολέ, να συζητήσουμε με του αρμοδίου επιτοπίω και να έχουμε μια πιο στενή παρακολούθηση μέσω αντιπροσωπιών τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Και εδώ επανέρχομαι στο σημείο εκκίνησης για το πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινέ διαπιστώσει. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ του ποσοστού σφαλμάτων όπως αναφέρεται από το ελεκτικό συνέδριο και όπως την καταμετράτε εσείς ως Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Και δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα από τις απαντήσεις σας και τις διευκρινήσεις που μας έχετε δώσει πού βρίσκεται η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών. Θα θέλαμε να υπάρχει λοιπόν μια εξέλιξη όπου θα υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ Κομισιών και Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των σφαλμάτων και των ποσοστού σφαλμάτων, ώστε να έχουμε ένα κοινό έδαφος επί του οποίου μπορούμε να προχωρήσουμε για την μείωση των σφαλμάτων. Σε άλλες γενικές διευθύνσεις τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Παραδείγματος χάρη στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης υπήρξε <clears throat> μία μεγάλη προσέγγιση μεταξύ Κομισιών και Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση των σφαλμάτων, κάτι το οποίο μας δίνει πιο ένα, ένα πιο ασφαλές έδαφος για να παρακολουθούμε τα θέματα αυτά. Μας είπε το Ελεκτικό Συνέδριο ότι οι στατιστικές οι οποίες δίδονται από τα κράτη-μέλη είναι πολλές φορές αναξιόπιστες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πρέπει να τροποποιηθεί. Και ενδεχομένως χρειάζονται περισσότεροι και πιο στεναρή λογιστική έλεγχη επιτόπου από την Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να τύχει της ε, αμέριστης προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών είναι αξιόπιστα και μας δίνουν μια ακριβή απεικόνηση της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ, ο κύριος Μπάρστας και ο κύριος Πίμπαλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την προσπάθεια την οποία έκαναν μέχρι τώρα. Να στραφώ τώρα προς τον κύριο Τσίολος και τις υπηρεσίες του. Νομίζω ότι απάντησαν ε, με αρκετά πλήρη τρόπο στις ερωτήσεις τις συμπληρωματικές οι οποίες έχουν τεθεί από πλευρά του συνεδρίου. Ένας από τους ελεγκτές του συνεδρίου είπε ότι τα στοιχεία και οι συγκρίσεις πρέπει να γίνουν με τα αποτελέσματα του παρελθόντος για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σωστή κρίση. Δύο διδάγματα νομίζω από όλα αυτά ε, βγαίνουν για μας. Καταρχάς, Αυτά τα οποία γνωρίζαμε τώρα είναι προσδιορισμένα ρυθμητικά. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο αναφέρεται περίπου στο 15% του συνόλου των πληρωμών. 0,4% των εποφελουμένων παίρνουν άνω των 100.000 ευρώ, δηλαδή το 11%. Αυτά όλα τα υποθέταμε, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι επιβεβαιωμένοι αριθμοί και ποσοστά. Μπορείτε λοιπόν κύριε Επίτροπε περαιτέρω να μας εξηγήσετε σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πού βρίσκεστε στις διαπραγματεύσεις σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις αυτές στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Ε, ακολουθούν θα έλεγα τις δικές σας κατευθύνσεις έτσι ώστε το 4% των γεωργών να μην παίρνουν το 11% του προϋπολογισμού, ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να μην παίρνει παρά το 15%. Ένα δεύτερο στοιχείο συνδέεται με την έννοια, με τον ορισμό μάλλον, του ε, ενεργού γεωργού. Υπάρχει και ο γεωργός του καναπέ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη διαφοροποίηση. Εδώ στην ουσία πηγαίνουμε προς τον καθορισμό ενός αρνητικού καταλόγου. Υπάρχουν αεροδρόμια, υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι, υπάρχουν αισιοδρομικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερα γεωργική δραστηριότητα και δεν θα πρέπει να εντάσσονται στο προβλεπόμενο σύστημα. Αλλά ποιος είναι πραγματικά ο δραστήριος, ο ενεργεία γεωργός αυτός ο ορισμός του ενεργεία γεωργού είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν υποτίθεται τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι στην ουσία θα ξαναγυρίσουμε στις αμαρτίες του παρελθόντος. Θα υπάρξουν δηλαδή ορισμένες προσπάθειες ορισμού στα πλαίσια των οποίων τα κράτη-μέλη δεν θα αντιμετωπίζουν ισότιμα τους γεωργούς και κάποιοι μάλιστα μη γεωργοί θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σάλτσο, κύριε Σπίφα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, το Ελεκτικό Συνέδριο για την πλήρη και θετική πληροφόρηση που μας έδωσαν. Θα ήθελα τώρα να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν ένα βασικό για μένα ερώτημα που έχει να κάνει με την επόμενη περίοδο προγραμματισμού στον επόμενο δημοσιονομική περίοδο για τον πρώτο πυλώνα της αγροτικής πολιτικής έχουμε μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία πολλαπλή συμμόρφωσης. <clears throat> έχουμε περισσότερες ε, ε, απαιτήσει για τα θέματα του περιβάλλοντος από ό,τι, θα, από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Και τώρα το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε εσεί ότι δεν θα προκύψει και ένα υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων από τις μεγαλύτερε απαιτήσει συμμόρφωσης, γιατί σε πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της υψηλή γραφειοκρατίας και των πολλών σφαλμάτων, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να απομακρυνθούν από το ευρωπαϊκό σύστημα πολλαπλή συμμόρφωση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η δράση τη Κομισιόν για να μπορέσει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων ότι θα περιοριστεί ο αριθμός των σφαλμάτων και των ποσοστώτων. Το δεύτερο ερώτημα είναι ίσως ε, υποδέστερο σε σχέση με το πρώτο ερώτημα. Πρόκειται για τα μέτρα χρηματοδότησης, ιδίως της αγροτικής ανάπτυξης και ξέρω ότι στον τομέα αυτό πολλές φορές τα κρατη έχουν δημιουργήσει τα ίδια πάρα πολύ πολύπλοκους κανόνες και αυτό έχει εντοπιστεί και από το ελεκτικό συνέδριο διότι θεωρεί ότι αυτοί οι κανόνες, οι πολύπλοκοι κανόνες δεν τηρούνται στην πράξη <clears throat> πάντοτε. Στη δική μου περιοχή βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ενόχληση και διαμαρτυρία των γεωργών για τα θέματα της γραφειοκρατίας γιατί οι κανόνες εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο με πολύ πολύπλοκο τρόπο. Τι μπορεί να κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πει «Μα δεν μπορείτε να θεσπίζετε τόσο πολύπλοκους κανόνες». Σας παρακαλώ να έχετε απλούστερους κανόνες. Έχετε λοιπόν το δικαίωμα παρέμβασης για να επιβάλλετε την απλοποίηση των κανόνων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για μένα. Και φυσικά ενδιαφέρει και τους γεωργούς. Και το, το επόμενο με ερώτημα είναι το εξής. Είναι για το ποσοστό επανίσπραξης των ποσών αυτών που είναι αντικείμενα σφαλμάτων. Για ορισμένε χώρε είχαμε θετικά αποτελέσματα. Αλλού όχι. Είχαμε αυτόν τον κανόνα του 50-50%. Αλλά για μένα το ερώτημα για τον προπολογισμό του 2011 είναι πώς κρίνεται την εφαρμογή αυτού του κανόνα 50-50% είναι μια επιτυχία η εφαρμογή αυτού του κανόνα. Και σε σχέση με τον κανόνα του 100% δηλαδή ότι πρέπει να απαιτηθεί αυτό το ποσό από το, από, στο σύνολό του από τον εθνικό προϋπολογισμό μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια ρήτρα. Θα δεχτούν τα κράτη-μέλη να ανακτάτε το ποσό το οποίο α, α, οφείλεται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς ή όχι. <clears throat> Και το τελευταίο μου ερώτημα. Και τώρα το θέμα που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των αγροτεμαχίων. Και πρόκειται για το θέμα των επιδοτήσεων που δίδονται σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες δεν είναι ακριβώς γεωργικού χαρακτήρα. Και έχετε πει ότι θα προχωρήσετε σε κάποιες μορφές έλεγχου. Το ερώτημά μου είναι αυτό βρίσκεται μέσα στις ηλικίε δυνατότητες της Κομισιόν να παρέμβει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι αυτό ο έλεγχος θα μπορέσει να γίνει αποτελεσματικά και θα υπάρξει μια αποτελεσματική παρακολούθηση ή έχετε την εμπιστοσύνη στα κρατημέλη ότι θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στα ίδια τα κρατημέλη αυτόν τον έλεγχο. Έχετε κάποιες ε, πραγματογνωμοσύνες σε σχέση με το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η παρακολούθηση. Αυτά λοιπόν από τη δική μου πλευρά και από την πλευρά του ΕΛΚ. Ο κύριος Μούλντερ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Ελεκτρικού Συνεδρίου και τον Επίτροπο για το φετινό τους έργο και η γενική εντύπωση που αποκομίζει κανείς είναι ότι όλοι χαρακτηρίζονται από τι καλύτερε δυνατές προθέσεις. Καλό είναι αυτό. Όλοι θέλουν να βελτιωθούν τα πράγματα, ποτέ δεν βελτιώνονται όμως στην πράξη. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο Μιλάμε για 18 χρόνια για το πολιτισμό σε νομικό πλαίσιο. Ποτέ δεν μα έδωσε μια θετική δήλωση το ελληνικό συνέδριο. Μα τέλο πάντων τι κακό συμβαίνει στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το ίδιο θυμοτυπικό έχουμε κάθε χρόνο. Και αν δει κανεί ε, τον τρόπο, τον πληρέστη, το διεξοδικότατο με τον οποίο απάντησε στο Κοινοβούλιο Κομισιόν, δεν έχω να πω ε, πάρα πολλά πράγματα. Φαίνονται να είναι όλα καλά. Μόνο στο τέλο το βλέπουμε ότι δεν ήταν τελικά τόσο καλά όσο φαίνονταν στην αρχή τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει μας εδώ στο Εκνοβούλιο. Η Ναυαρχίδα, αν θέλετε, της, του δημοσιονομικού ελέγχου ήταν το σύστημα Άγιαξ, ο ΕΑΣ, και θέλαμε να είμαστε κάτω από το 2% του ποσοστού σφάλματος, πάλι το έχουμε υπερβεί και αυτό πραγματικά μας ε, ενοχλεί ιδιαίτερα. Πάλι κάτι δεν πήγε καλά, ενώ λέγαμε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Εντάξει, μπορούμε να προσθέσουμε νέες προποθέσει, ε, νέους όρου κτλ. Αλλά γιατί ένα σύστημα που κάποτε λειτουργούσε καλά τα επόμενα διαδοχικά χρόνια επιδεινώνεται. Πού οφείλεται αυτό. Στο Κοινοβούλιο είχαμε σκεφτεί ως λύση ότι μπορούμε να κάνουμε πολλούς ελέγχους και νομίζω ότι πολλοί, πολλοί αγρότες για παράδειγμα στην Ευρώπη έχουν μπουχτίσει πια. Δεν αντέχουν άλλους ελέγχους. Του ελέγχει το συνέδριο, οι κομισιόν, ε, του ελέγχουν εθνικέ κυβερνήσεις, ε, οι περιφερειακέ όπου υπάρχουν κτλ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τον ιδιωτικό κλάδο, την ιδιωτική μηχανή που και αυτή ελέγχει. Γιατί κάποιο δεν παραδίδει μόνο το γάλα, το παραδίδει υπό συγκεκριμένου όρου και προποθέσει. Και ούτω Υπάρχουν λοιπόν ε, συστήματα ελέγχου και για την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων αλλά είναι κάτι που δεν το βλέπουμε αλλού στον κόσμο, χωρίς όμως παρόλα αυτά να μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τα συστήματα. Εμείς θεωρούμε ότι η Κομισιόν έχει την πολιτική ευθύνη και πιστεύουμε ότι θα πρέπει και αυτή από την πλευρά της να καταστήσει υπεύθυνα τα κρατη Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή θέλουμε να υπάρξει πολιτική ευθύνη για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Διότι εάν ζητήσουμε δήλωση ε, στο τέλος του χρόνου για, στα μέλη, από κάποιον πολιτικό υπεύθυνο και αν αυτός ή αυτή είναι στην ίδια θέση με την Κομισιόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για την πολιτική υγεία, αν θέλετε, αυτού του ατόμου στη συγκεκριμένη χώρα μέλος. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν καλό να προχωρήσουμε. Και έχω και δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη, αν δείτε την έκθεση, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι γεωργικών επιδοτήσεων που κατονομάζονται τις απαντήσεις κομισιών, κάποιοι από αυτούς είναι κρατικές επιχειρήσεις από τα νέα κρατημέλη. Κατά την άποψη της Κομισιών, αιτιολογείται αυτό, είναι δικαιολογημένο. Γιατί κατά την άποψή μου αυτό υπερβαίνει του στόχου τη κοινή γεωργικής πολιτική. Θα πρέπει να είναι επιδότηση, θα πρέπει η επιδότηση να πηγαίνει σε μεμονωμένου παραγωγού. Τι πιστεύει σχετικά λοιπόν η Κομισιόν. Σω θα ήταν δυνατόν να γίνουν κάποιε αλλαγέ στον νέο κανονισμό για τη γεωργία. Αλλά είναι δικαιολογημένο αυτέ οι κρατικέ, αυτοί οι κρατικοί φορείς να λαμβάνουν επιδοτήσει. Και κάτι άλλο που δεν έχω δει βέβαια σε κάποια έκθεση, αλλά το θυμάμαι από προηγούμενε χρονιέ όταν αλλάζαμε την κοινή γεωργική πολιτική και είχαμε την ε, ενίσχυση εισοδήματο σε ό,τι αφορά την διοκτησία. Εκεί βασίζονταν στην διοκτησία των γεών. Και πάντα μιλούσαμε για την Ελλάδα που δεν έχει χρηματολόγιο. Παρ' όλα αυτά παίρνανε τις ε, πληρωμές οι αγρότες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο, γιατί δεν ξέρεις ποιος ε, είναι ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου, πώς δίνεις τις συνεισίες. Έχω διαβάσει διάφορα άρθρα ε, για την Ελλάδα και ξαναδιαβάζω και τώρα. Υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή ειδικών που βρίσκεται στην Ελλάδα και η οποία βοηθά και σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο, το σύστημα καταγραφή των αγροτεμαχίων. Πώ λοιπόν έχει κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα, θα ήθελα να μα πει η Κομισιόν. Τι πληροφορίε έχει, ευχαριστώ. Πολλέ ερωτήσει, λέει ο Πρόεδρο. Περνάει ο χρόνο όμω, πετώντα. Έχω άλλου τρει συναδέλφου και μετά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Κύριε κυρία Ανδρέα είναι επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στο ελεκτικό συνέδριο. Ο κύριος Κούμπικ είπε στα σχολιά του ότι θα πρέπει να περιμένουμε πολλά χρόνια για να δούμε για να δούμε αν υπάρχει πράγματι στατιστική τάση ή όχι. έχουμε αύξηση πραγματικούς όρους ε, τη τάξη του 1,5%. Αν έχουμε συνεχόμενα αυξήσεις λοιπόν σε γενικού όρους, ε, για οποιονδήποτε βλέπει ε, την επιτυχία, αν θέλετε, ή μη επιτυχία των πολιτικών, διαπιστώνει ότι δεν είναι αξιόπιστος ο έλεγχος των πολιτικών. Άρα το ερώτημα που έχω προς το ελληνικό συνέδριο είναι πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν υπάρχει τάση ή όχι. Μα υπάρχει ήδη ιστορικό ποσοστό σφαλμάτων. Δώστε μας λοιπόν ε, μία απάντηση. Πόσα χρόνια ακόμα πρέπει να περιμένουμε. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να πούμε ότι ναι πράγματι υπάρχει αυτή η τάση. Επίσης τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής. Άρα είναι πολύ σημαντικό τις αποφάσεις μας να τις βασίσουμε και στο παρελθόν. Από τον Επίτροπο Τσιόλος, ο οποίος παραδέχεται ότι δεν είναι ικανοποιητικό αυτό το ποσοστό σφάλματος, ε, και λίγα λέτε κατά την άποψή μου, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Αλλά λέτε επίσης, κύριε Τσιόλος, ότι αυτό δεν συνιστά και απάτη ή λέτε ότι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα ποσά αυτά που έχουν χαθεί. Σε μια από τι απαντήσει σα λέτε ότι σε περίπτωση που η ότι δεν γίνεται με τη δεύτερη επιμέλεια η ανάκτηση, τα μία ποσά θα χρεωθούν στους εθνικούς περιπολογισμούς των κρατών μελών. Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη είναι σε θέση τώρα, αυτή τη στιγμή, με την κρίση αυτή, με τα μέτρα λιτότητας, να αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση, δηλαδή με χρήματα των φορολογουμένων ακόμη περισσότερα μπορέσουν να σταθμίσουν τα διαφυγόντα αυτά ε, ποσά. Και τώρα σε ό,τι αφορά τη δήλωση για τις επιλέξιμες περιοχές. Τώρα, αυτό είναι απάτη ή δεν είναι, κατά την δική σας άποψη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Je donne la parole à Jean-Pierre Audi. Merci, Monsieur le, Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τις εξηγήσεις του. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για τα γαλλικά σας. Κάθε φορά που παραβιάζονται οι αρχές της πολυγλωσσίας κάνω ορισμένε παρατηρήσεις γι' αυτό. Και όταν είχαμε περάσει το δημοσιονομικό έγγραφο των 400 σελίδων θυμάμαι ότι <clears throat> δεν ήταν σε όλες τις γλώσσες διαθέσιμο. Εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε κάτω από την πίεση του χρονοδιαγράμματος και δύσκολα θα εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας, φτάνοντας το 13, ότι βιαζόμαστε, ενώ στην ουσία ασχολούμεθα με αριθμούς του 2011. Τον Απρίλιο στην ουσία εμείς θα κληθούμε να ψηφίσουμε κάποιες παρατηρήσεις ε, ε, χωρίς να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τα διορθωτικά στοιχεία τα οποία έχουμε ανάγκη για το μέλλον ιδιαίτερα στα πλαίσια της ψηφοφορίας όλων των εγγράφων, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την προγραμματική περίοδο 14-20. Στο χαρτοφυλάκιο για το οποίο είστε υπεύθυνο, κύριε Επίτροπε, ε, πόσες πιστώσεις πηγαίνουν σε τελικούς χρήστες. Θέτω το ερώτημα αυτό στους επιτρόπους τους οποίους ε, δεχόμαστε, γιατί διαρωτώ με αν η δειγματοληψία ε, της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου που είναι 180 στην γεωργία και 160 στην ανάπτυξη της υπαίθρου θα ήθελα πως ε, επί τη βάση ενός δείγματος 180 πληρωμών βρίσκει 39% λαθών και στο τέλος λέει ότι το λάθος όμως είναι 2,9%. Εγώ μεθοδολογικά δεν το κατανοώ αυτό, δεν κατανοώ την τεχνική αλληλουχία, και θα ήθελα να ζητήσω από το συνέδριο με ένα επεξηγηματικό σπνημόνιο για το πώς φτάνει στο 2,9 ενώ ανοιχνεύει στα 180-39%. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω και το σύνολο των ποσών που καλύπτονται από τις πληρωμές αυτές και άκουσα με ανησυχία τον κύριο Κούμπικ, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στα ποσοστά λαθών, ότι η ποιότητα της προσπάθειας των πιστοποιητικών αρχών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτή με επιφυλακτικότητα και ότι οι αρχές πληρωμών λειτουργούν με πάρα πολλές ελλείψεις ακρίβειας. Τώρα για το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι παρόν στη συνεδρίασή μας, δεν ξέρω αν θα του δώσετε το λόγο. Στις ανταλλαγές απόψεων που είχαμε εμείς μέχρι τώρα όμως αμφισβητούμε ουσιαστικά τη συμπεριφορά των κρατών μελών. Περιπλέκουν τα πράγματα περισσότερο. Διαχειρίζονται το μεικτό αυτό επίπεδο διαχείρισης με πάρα πολύ υψηλά λάθη, γιατί βασική υπεύθυνη είναι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και οι υπάλληλοι του. Δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για τα κράτη-μέλη, πρόκειται για εξωτερικές υπηρεσίες, πολιτικά αυτόνομες, και το Συμβούλιο όλων αυτό είναι ιδιαίτερα σιωπηλό. Δεν έρχεται στις ολομέλειές μας, δεν εκφράζει την άποψή του κτλ. Θα σας πει το Συμβούλιο ότι βέβαια δεν εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Πράγματι πρόκειται για έναν θεσμό sui generis. Δεν εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη γιατί τα κράτη-μέλη αυτό εκπροσωπούνται. Με ανεξάρτητο και αυτόνομο τρόπο. Παρόλα αυτά όμως σαν δεύτερη επί του προϋπολογισμού αρχή και σαν συνομοθέτη το Συμβούλιο καλείται να εκφέρει την άποψή του για τα θέματα των απαλλαγών γιατί έχει ένα τμήμα ευθύνη και αυτό στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια της αποκοινού διαχείρισης. Ε, Κύριε Επίτροπε, τώρα για σας κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι είναι ικανοποιητικό το ότι δεν υπάρχουν απάτες και ότι τα ποσά επί των οποίων υπήρχαν λάθη έδωσαν χώρο και σε κάποιες επιστροφές. Θα ήταν δυνατόν, διαρωτώ με, και αυτή είναι ερώτηση και για το ελεγκτικό συνέδριο. Ξέρετε ότι το 2014, πριν το τέλος της εντολής της δικής μας και της δικής σας, να μπορέσουμε κάτω από τεχνικές συνθήκες τις οποίες ακόμα αγνοώ ένα ποσοστό αξιολόγησης ε, για το σύνολο των λαθών από το 2007 μέχρι το 2013 δεν γίνεται βέβαια γιατί έτσι όπως δουλεύουμε εμείς το 2015 θα ξέρουμε τι έχει γίνει το 2013 αλλά εν πάση περιπτώσει μήπως μπορούμε να κατανείμουμε δημόσια προς τους εκλογείς μας μια αξιολόγηση συνολική και όχι μια ετήσια αξιολόγηση της οποίας ε, τα αδυναμίες γνωρίζουμε. 2007 λοιπόν ελεγχόμενη περίοδος μέχρι το 2011 ή 2012. Δεύτερη ερώτηση για το πρόγραμμα δράσης. Σας τέθηκαν ορισμένες γραπτές ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε πού βρίσκεστε σήμερα. Ποια θα είναι η χρησιμότητα αυτής της μεθόδου. Μια άλλη ερώτηση αφορά την απλοποίηση. Τέθηκε και από τον συνάδελφο Μίλντερ και από πολλούς άλλους βουλευτές. Οι πολίτες δεν μπορούν πια οι περιπλοκότητε, οι γραφειοκρατικές, εθνικές και κοινοτικέ είναι απαράδεκτες. Βλέπουμε και την άνοδο των ακραίων πολιτικών θέσεων. Εμείς οι δημοκράτες θα κάνουμε όλα δύσκολα. Και το ερώτημα το οποίο σας θέτω, που είναι λίγο εκτός θέματος βέβαια σχέση με την απαλλαγή, είναι ότι μιας και βρίσκεστε σε διαπραγμάτευση με τους συνομοθέτες για ένα σύνολο εγγράφων ε, για την επόμενη ε, περίοδο της ΚΑΠ μέχρι το 2020 σας δημιουργείται η εντύπωση ότι τα κοινοβούλια σαν παράδειγμα στην ουσία περιπλέκουν τα πράγματα και οι κυβερνήσεις το ίδιο ενώ η Κομισιόν έχει καταλάβει το πρόβλημα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι στο παρελθόν είχα την αίσθηση πριν λίγα χρόνια ότι ήταν ένας παράγων περιπλοκοποίησης σε εισαγωγικά η λέξη. Ενώ βλέπω τώρα ότι έχει κατανοήσει το πρόβλημα και προσπαθεί να τα απλουστεύσει. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δημιουργείται. Όταν διαβάζει κανείς την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πίνακες επιδόσεων της απλοποίησης ή απλούστευσης που έχουν ε, δημοσιευθεί, ε, εκπλήσωμε αρνητικά γιατί δεν βγάζουμε τα συμπεράσματα και τα διδάγματα από αυτά τα οποία συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια και στην ουσία δημιουργούμε, τροφοδοτούμε το αίσθημα το αντιευρωπαϊκό επί τη βάση της έλλειψης παρεμβάσεών μας στο συγκεκριμένο θέμα σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών. Ευχαριστώ, ο Μάρτιν Χόισλιν. Κάποια σύντομα ερωτήματα προς τον Επίτροπο και το Ελεκτικό Συνέδριο. Πολλές φορές υπήρξε, υπήρξαν πολλά προβλήματα με τις χορτολιβαδικές ε, εκτάσεις. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είδαμε και στη συζήτηση για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Τι ακριβώς είναι μια χορτολιβαδική έκταση. Και το συζητήσαμε αυτό το θέμα πολλές φορές με την Επιτροπή Γεωργίας, παραδείγματος χάρη στην περιοχή των Άλπαιων στην Αυστρία, να δούμε πώς μπορεί να διαχωρίσουμε μια αλπική περιοχή από μια άλλη περιοχή που έχει διαφορετικά είδη Είναι λοιπόν κύριε Επίτροπε ένα θέμα συγκεκριμένου ορισμού το τι είναι μια, ε, ένας λιμόνας, μια χορτολιβαδική περιοχή και επίσης υπάρχει το θέμα του ελέγχου της διαδικασίας πιστοποίησης. Άμα δεν λειτουργεί σωστά αυτή η διαδικασία της πιστοποίησης θα έχουμε προβλήματα. για τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία και αυτά παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό σφαλμάτων. Είναι βέβαια ένα πρόβλημα με τη νέα διαμόρφωση που παίρνει η αγροτική πολιτική. Αν αυτά τα νέα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα είναι τόσο επιβαρυντικά για τον Γεωργό και έχουν να κάνουν με, το λεγόμενο πρασίνισμα της Γεωργίας και βλέπουμε ότι έχουν τόσα πολλά προβλήματα μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εφαρμογής της κρατικής πολιτικής ή θα θέλαμε να έχουμε τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν αυτόματα σαν greening, σαν μέτρα πασινίσματος της γεωργίας, ορισμένες μορφές χρήσης των ε, αγροτεμαχίων. Επομένως, πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν τα υψηλά ποσοστά ασφαλμάτων που έχουμε δει σε επίπεδο μέτρων περιβάλλοντος. Και εγώ επίσης θα συμφωνήσω με τον κύριο τον κύριο Γκάιερ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατονομαστούν και τα κράτη τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων. Έχουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών, τελικά πληρώνει την ύφη συνολικά η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόνται τα προβλήματα. Επίση το ερώτημα του τι είναι ενεργός γεωργός. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Γεωργίας. Δεν είναι καθόλου απλό να βρούμε ένα συγκεκριμένο ορισμό για τι αποτελεί ενεργό γεωργό. Μπορούμε να θέσουμε ένα όριο οικονομικών δραστηριοτήτων, ένα όριο τζίρου για το γεωργό, αλλά πολλές φορές ξέρουμε ότι ένας γεωργός μπορεί να ασκεί και άλλες δραστηριότητες, είτε ερασιτεχνικά, είτε για άλλους λόγους και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ένα ενιαίο ορισμό για την ενεργή δραστηριότητα του κυρίου Γεωργού. και επίσης για τις κρατικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουμε και κάποιο ανώτατο όριο για τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Μάρτιν. Και τώρα. Κύριε Επίτροπε, είχατε ένα ευρύ πεδίο ερωτήσεων και είναι η ευκαιρία να απαντήσετε σε όλα αυτά τα πολλαπλά ερωτήματα, κύριε Επίτροπε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για τον ε, εισηγητή, για τον κύριο Γκάγερ. Ακούστε, σε ό,τι αφορά την γενική εκτίμηση του ελεγκτικού συνεδρίου, όπως είπα στην παρέμβασή μου, για τον πρώτο πυλώνα, η εκτίμησή μου, όπως ε, αυτή και του κύριου Κούμπικ, είναι ότι είμαστε μέσα στην ψαλίδα αυτή της διακύμανσης ε, των λαθών που τα τελευταία χρόνια δεν έχει παρουσιάσει σημαντική διαφορά. Αν συγκρίνουμε πολύ απλά το μέσο ποσοστό, το πλέον πιθανό μέσο όρο σφαλμάτων όπως τον αποκαλούμε, βλέπουμε κάποιες δεκιμάνσεις. Η μεθοδολογία όμως από στατιστικής πλευράς είναι τέτοια που δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ποιος είναι ακριβώς ο συντελεστής σφαλμάτων. Έχουμε λοιπόν αυτή την ε, λίγο πολύ ίδια, παρόμοια διακύμανση. Αυτό απαντά και το ερώτημα της κυρίας Ανδρέας. Γι' αυτό και είπα ότι από συστημική πλευρά, λόγω του συστήματο που έχουμε, το ΝΕΑΝΤΑ, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση ελέγχου, αυτή τη βάση δεδομένων, αυτό το σύστημα μα δίνει δυνατότητα να κάνουμε διαχείριση των πραγμάτων. Αν όμω υπάρχει καλή ε, συντήρηση και διατήρηση των βάσεων δεδομένων. Δεν έχουμε συστημικό πρόβλημα της αξίας, της ποιότητας του συστήματος, αλλά το θέμα είναι πώς το συντηρούμε, το διατηρούμε το σύστημα για να έχουμε αποτελεσματικά δεδομένα. Αυτό που διαπιστώσαμε, όπως και το συνέδριο βέβαια, είναι ότι σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γενικό πρόβλημα, τουλάχιστον κατά τη δική μας εκτίμηση, σε ορισμένα λοιπόν κράτη-μέλη, συνεχίζεται να παρουσιάζεται ακριβώς πρόβλημα με την ποιότητα των δεδομένων της βάσης δεδομένων για τα αγροτεμάχια, πώς μετρώνται και η βάση δεδομένων με τους εργούς τους αγρότες. Αλλά τα αγροτεμάχια τώρα και εντοπισμό των επιφανειών, των επιλέξεων επιφανειών, εκεί μπαίνει το θέμα. Έχουμε κράτη-μέλη που έχουν καλύτερη βάση δεδομένων πάλι. Υπάρχουν ε, χώρες, γιατί ρωτήσατε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα λοιπόν πράγματι υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα τις προηγούμενες χρονιές. Υπήρξαν σχέδια δράσης όπου η Ελλάδα ακόμη και δεν είχε κτηματολόγιο που είναι μια νομική βάση δεδομένων, έχει εκπονήσει μια βάση δεδομένων με τα αγροτεμάχια που ορίζονται, οριοθετούνται. Άρα τώρα μπορούμε κάπως καλύτερα να εντοπίσουμε τα ασφαλότητα. Σίγουρα μακρόπνο αυτό το έργο, πάντως υπάρχει εντοπισμός, υπάρχει ταυτοποίηση αγροτεμαχίων, είναι πιο σταθερά τώρα πια. Σε άλλα κράτη-μέλη δεν μπορούμε να πάμε σε επίπεδο αγροτεμαχίων, αλλά ε, σε, στα λεγόμενα φυσικά μπλοκ. Εκεί μπορεί να υπάρχουν από μια χρονιά στην άλλη προβλήματα για το πώς οι οριοθετούν τα αγροτεμάχια. 24 εκτάρια ραβοσίτου τη μια χρονιά, μετά σίτου και δεν ξέρω εγώ τι. Ε, υπάρχει κάποια μετακίνηση, κινητικότητα, πώς να το πω, των αγροτεμαχίων. Εδώ δεν είναι συστημικό βέβαια το πρόβλημα, αλλά ποιότητα δεδομένων. Και εκεί πρέπει να δώσουμε την προσοχή. Και το θέμα των πληροφοριακών συστημάτων είναι θέμα. Τώρα μηχανογραφείται ε, σε πολλές χώρες ε, η και, και η διαδικασία καταβολή πληρωμών και μπαίνουν και κάποια στοιχεία στη βάση δεδομένων. Αλλά σε ό,τι αφορά τη διόρθωση των στοιχείων, σε κάποιε περιπτώσει δεν γίνεται καλή δουλειά. Αλλά με του ελέγχου μα μπορούμε να βρούμε τα προβλήματα στον τομέα αυτό. Και ιδίω με την εκαθάριση των λογαριασμών και τη συμμόρφωση, έχουμε συστήματα χρηματοοικονομική διόρθωση που αποθαρρύνουν τα κράτη-μέλη από το να μην προσέξουν αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, τα ενθαρρύνουμε, για να το πω με να προσέχουν. Γιατί αν δεν εντοπιστούν τα προβλήματα αυτά, θα πληρώσουν τα κρατη για αυτές τις διορθώσεις ε, και εποφελούμε τις ε, ευκαιρίες για να απαντήσω στην κυρία Ρέσεν που λέει γιατί πρέπει τις διορθώσεις να πληρώσουν τα κρατη Ακούστε γιατί. Είμαστε στην ε, μεικτή διαχείριση. Δεν είναι δικά μας χρήματα, δεν είναι χρήματα της Κομισιόν, είναι χρήματα των κρατών μελών. Αν λοιπόν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν εσφαλμένως τα χρήματα αυτά και αν οι εθνικές διοικήσεις δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, πρέπει να αναλάβουν την οικονομική ευθύνη γιατί είναι χρήματα των φορολογουμένων. Και αυτά που δίνονται και αυτά που δαπανώνται. Τα ίδια χρήματα είναι τα χρήματα των φορολογουμένων. Απλά είναι σε ποια κολόνα, σε ποια στήλη τα βάζουμε. Έχουμε λοιπόν ζήτημα διαχείριση. Εμεί αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα, αλλά σε ό,τι αφορά αυτή την κοινή μεικτή διαχείριση, όταν έχουμε πρόβλημα σε επίπεδο κρατομέλων, πρέπει και αυτά τα κρατημέλη δηλαδή να αναλάβουν τι ευθύνε του και δεν μπορούμε επαόριστο να αυξάνουν τον αριθμό των ηλεκτών τη Κομισιόν για να κάνουμε εμεί τη δουλειά των 27 κρατών μελών. σω αυτό να ήταν πιο εφικτό πριν από 20 χρόνια που ήταν λιγότερα τα κρατημέλη. Τώρα όμω πια δεν είναι δυνατόν. Άρα αυτή η μεικτή διαχείριση, κοινή διαχείριση πρέπει να λειτουργήσει. Και τώρα θέλω να επανέλθω στο σχέδιο δράση. στα σχέδια δράσης, δηλαδή το δεύτερο πυλώνα ανάπτυξη τη υπαίθρου όπου το ποσοστό ε, σφαλμάτων είναι πιο υψηλό. Η πρώτη μας ανάλυση δείχνει ότι αυτό οφείλεται και στην ποιότητα των ελέγχων που διεξάγονται επί τόπου τώρα, ποιότητα ελέγχων, δηλαδή ποιότητα προσωπικού, αλλά και σαφήνεια για το έργο του ελεγκτή επιτόπου. Και δεύτερος λόγος, πολυπλοκότητα του προγραμματισμού, δηλαδή πώς χρησιμοποιούνται από τα κρατημέλη τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κριτήρια επιλογής, εσμεύσεις από τους αγρότες. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά το συζήτησα με τον κύριο Γκάγερ και όλα αυτά θα τα συμπεριλάβουμε στο σχέδιο δράσης το οποίο θα προτείνουμε να εφαρμοστεί και μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει εφαρμογή. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των ελέγχων, αλλά και από την άλλη πλευρά στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους, για να δούμε, να εντοπίσουμε καλύτερα πού ε, βρίσκουμε προβλήματα, πού υπάρχουν προβλήματα με τους έλεγχους. Και επίσης, δεύτερο στοιχείο, απλούστευση των προγραμμάτων. Και μπορεί, ε, αυτό μπορεί να γίνει και τώρα για τα προγράμματα που ήδη τρέχουν, και πρέπει βέβαια εκεί να δώσουμε προσοχή στο περιεχόμενο και στην δυνατότητα ελέγχου, στην ελεγξιμότητα αν θέλετε, αλλά και για την επόμενη χρήση, για τον επόμενο μεσονικό έτος βλέπουμε θα δούμε όταν εγκρίνουμε προγράμματα όχι μόνο την ε, πολιτική βιωσιμότητα των πολιτικών στόχων δηλαδή πρέπει να επιτευχθούν από το πρόγραμμα αλλά και την ελεγξιμότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων. Αυτό θα πρέπει να συμβαδίζουν και θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ του στόχου της επίτευξης αποτελεσμάτων πολιτικά, οικονομικά κτλ. Αλλά όχι με κάθε τίμημα. Ναι, με να υπάρχουν αποτελέσματα, αλλά να δείξουμε ότι και τα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι και αυτά διαφανή, ξεκάθαρα και ελέγξιμα καλύτερα. Αυτά τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων τώρα τα εντοπίζουμε γιατί, γιατί αυτό έρχεται σε ποια κράτη-μέλη. Σε 14 περίπου κράτη-μέλη με τα οποία και συνεργαζόμαστε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ή δύο κράτη-μέλη. Φυσικά, εγώ έχω εδώ τον κατάλογο μπροστά μου. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σα ε, είναι χρήσιμο, αλλά έχουμε την Αυστρία, τη Δανία, την Εστονία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Λετωνία. Σε αυτές τις χώρες είναι υψηλότερα τα ποσοστά ασφαλμάτων γιατί είναι πιο πολύπλοκα και τα προγράμματα. Άρα είναι και θέμα προσέγγισης των κρατών μέλων αυτών. Επειδή όμως θεωρούμε ότι είναι ήδη τα μισα κρατημέλη, άρα το πρόβλημα αυτό είναι μάλλον γενικό. Άρα πρέπει να δούμε και το ζήτημα της πολυπλοκότητας των προγραμμάτων γενικότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα των ελέγχων, εκεί όπου βλέπουμε να υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα ή άλλο κράτος μέλος, έχουμε και ειδικά σχέδια δράσης με τα λογω κράτη-μέλη για το ζήτημα της ποιότητας των ελέγχων συγκεκριμένα. Τώρα, πώς θα καταρτήσουμε μια λειτουργική βάση, γιατί έχουμε διαφορά μεταξύ εκτιμήσεων του συνεδρίου και δικών μας εκτιμήσεων. Δύο ε, στοιχεία ως εξήγηση μπορώ να σας δώσω. Πρώτα απ' όλα, οι ε, αναλύσεις του συνεδρίου, του ελεκτρικού συνεδρίου, βασίζονται σε ένα σύστημα δειγματοληψίας, που είναι για το συνέδριο ειδικά, ε, το έχει εξηγήσει γιατί το χρησιμοποιεί το συνέδριο δεν μπορεί να κάνει όσου ελέγχου μπορούμε να κάνουμε εμεί, άρα κάνει δειγματοληψία. Εμεί, Ω Κομισιόν βασίζουμε τι αναλύσει μα σε ελέγχου που διενεργούνται από τα κράτη-μέλη, αλλά και σε ελέγχου που διενεργούμε εμεί για την ποιότητα των ελέγχων των κρατών μελών. Για να απαντήσω και στο ερώτημα του κυρίου Οντί, για τον πρώτο πυλώνα, 10 εκατομμύρια περίπου είναι δικαιούχοι. 10 εκατομμύρια πράξεις δηλαδή περίπου έχουμε και έχουμε λίγο πολύ 500.000 ελέγχους, λίγο παραπάνω 500.000 ελέγχους. Για τις άμεσες πληρωμές έχουμε και διοικητικό έλεγχο επί του συνόλου των πράξεων των συναλλαγών. Περίπου λοιπόν 500.000, 580.000 έλεγχοι επιτόπου. Για το δεύτερο πυλώνα, 5,7 εκατομμύρια συναλλαγών πράξεων έχουμε, τόσους δικαιούχους δηλαδή, και εκεί περίπου 500.000 ελέγχους έχουμε πραγματοποιήσει, μάλλον έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη-μέλη. Ο αριθμό των ελέγχων είναι σημαντικός, γιατί βάσει του αριθμού των ελέγχων και βάσει των ελέγχων υπολογίζεται από την Κομισιόν και το διάστημα και ε, των σφαλμάτων και το πλέον πιθανό λάθος. Και έχουμε ουσιαστικά ε, σφάλματα αλλά και σφάλματα διαδικαστικά που δεν επηρεάζουν όμως τελικά Γι' αυτό είπα, άλλο είναι το σφάλμα και άλλο είναι κατά πόσον θα γίνει κακή χρήση των πόρων ή θα χαθούν κάποια χρήματα στο πλαίσιο του τελικού στόχου. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, Παραδείγματος διαγωνισμός για έργα οδοπίας. Ε, αν υπάρχει ένα σφάλμα, ακόμη και αν είναι 100%. Αν ο δικαιούς δηλαδή δεν έχει σεβαστεί όλους τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων για τη δημοσίευση του διαγωνισμού και για όλους τους κανόνες. Παρ' όλα αυτά προέβη στην επιλογή αναδόχου. Ο εργολάβος αυτός ε, έκανε τα έργα οδοποιίας. Έχουμε λοιπόν ε, εκτέλεση, δεν έχουν όμως γίνει σεβαστές οι διαδικασίες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι 100% αλλά είναι απάτη αυτό, δεν είναι. Ούτε είναι μη χρήση τελικά, μη αξιοποίηση των πόρων. Για όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν στην Κομισιόν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και τη δική μας ανάλυση για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων των κρατών μελών με στόχο να ενισχύσουμε τον ρόλο των φορέων πιστοποίησης. Στον Μουσιακό Κανονισμό για το επόμενο έτος, το οικονομικό, προτείνουμε πλέον συστηματικά οι οργανισμοί, οι φορείς πιστοποίησης να ε, εκτελούν με έναν προσωπευτικό μα σε κάθε κράτος μέλος ε, κάποιες αναλύσεις για να δούμε την ποιότητα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει οι οργανισμοί πληρωμών. Βέβαια, το ελεγκτικό συνέδριο ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά την ποιότητα του έργου των ε, φορέων πιστοποίηση. Σα υπενθυμίζω όμω ότι τώρα έχουμε ένα εθελοντικό σύστημα. Τι θα πει αυτό, αν τα κρατημέλη, αν οι φορεί πιστοποίηση αφισβητήσουν μια χρηματοοικονομική συναλλαγή, flat rate παραδείγματο χάρη που προτείνει η Κομισιόν, εκεί υπάρχει δυνατότητα δημιουργία ενό νέου αντιπροσωπευτικού δείγματο και υποβολή τη σχετική ανάλυση στην Κομισιόν, που και αυτή όμω κάνει ανάλυση. Αν θεωρούμε ότι δεν είναι ποιοτική δουλειά, δεν αναγνωρίζουμε το εθελοντικό αυτό έργο, την εθελοντική αυτή δουλειά για τη μείωση Θέλουμε όμως να είναι υποχρεωτικό αυτό από το 2014 και μετά, άρα θα δώσουμε κατευθυντήρες γραμμές. Θα δώσουμε αρχές πάνω στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η εργασία. Για να έχουμε ποιοτική ε, δουλειά από τους οργανισμούς πιστοποίησης, αφού θα υπάρχουν και πιο σαφείς κανόνες. Για την ενίσχυση λοιπόν των ελέγχων τώρα τη Κομισιόν των επιτόπιων ελέγχων και για την ενίσχυση των ρόλων των φορέων πιστοποίηση, θέλουμε να βελτιώσουμε και τα στατιστικά στοιχεία, την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που μας έρχονται από τα κράτη-μέλη. Είναι και αυτός ένας τρίτος στόχος για τον κύριο Μπεν Στάς, σε ό,τι αφορά τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε σε σχέση με τους δικαιούχους. Για να αριθμίσουμε το πρόβλημα, γιατί έχουμε ένα, μικρό, ένα μεγάλο αριθμό μικρών δικαιούχων και, μεγάλο, και μικρό αριθμό μεγάλων δικαιούχων εντό αγωγικών. Προτείνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να έχουμε ένα ανώτατο όριο για τι πληρωμέ που ξέρουμε ότι ουσιαστικά αποσκοπούν στη στήριξη του εισοδήματο και περιορίζεται στα 300.000 ευρώ για τους μεγάλους δικαιούχους. Ίσως όμως δυστυχώς το είδατε, το είδατε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο διαπραγματευτικό κουτί προτείνεται να είναι θελοντικό αυτό. Και αν είναι θελοντικό, δεν ξέρω πόσα κράτη-μέλη θα το εφαρμόσουν. Πάντως η Κομισιόν θα επιμείνει Ανώτατο όριο λοιπόν, επιβολή ανώτατων ορίων, που είναι η πρώτη λύση για να έχουμε ισότιμη κατανομή. Δεύτερον, εσωτερική σύγκληση των άμεσων πληρωμών σε επίπεδο κρατών μελών. Και εδώ έχουμε σημαντικέ διαφορέ εντό του ίδιου κράτου μέλου και μάλιστα και στην ίδια την περιφέρεια μεταξύ διαφορετικών εκμεταλλεύσεων. Αυτή λοιπόν η διαδικασία εσωτερική σύγκληση πιστεύω ότι θα μειώσει και αυτή, αυτό το χάσμα, αυτή τη διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρών δικαιούχων. Πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για τον κύριο Χόσλινγκ, Μπορεί να σα το πει. Στην κόμμα γκρι, αλλά και στο κοινοβούλιο είναι δύσκολε συζητήσει. Γιατί θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ισοτιμία και ισότητα. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι αρκετά απεσιόδοξο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το μέλλον τη επιβολή ανώτατου ορίου. Εμεί θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε βέβαια, αλλά προ το παρόν φαίνεται να μην, μας, να μην συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Ελπίζω πάντως να έχουμε με μια πιο σώτιμη κατανομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ενεργεία γεωργό, αγρότη, η Κομισιόν θα επιμείνει μέχρι τέλους να υπάρξει ευρωπαϊκός ορισμός. Να υπάρχουν δηλαδή ευρωπαϊκές αρχές και να υπάρχει μια αρνητική λίστα. Επίση, αφήνουμε και στα κράτη-μέλη ένα περιθώριο ευελιξία ώστε να προσθέσουν ενδεχομένω ειδικά κριτήρια. Τα κριτήρια όμω θα ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτά, τα κριτήρια που θα ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο, θα είναι Δεν θα είναι περιοριστικό ορισμό θα είναι προαιρετική συμπληρωματική ορισμοί από, από τα κράτη-μέλη. Για τον κύριο Πίπερ, αιρεσιμότητα περιβαλλοντική. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι για το πρασίνισμα η Κομισιόν θα αγωνιστεί μέχρι σε σχάτων για να παραμείνουν απλοί οι κανόνες και εύκολοι στον έλεγχο. Προτείνουμε εύκολους ως προς τον έλεγχο κανόνες, δηλαδή διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων, χρωτοδιβαλικών εκτάσεων. Έχουμε πολλά στοιχεία από τα κρατημέλη. Διαφοροποίηση καλλιεργιών. Εκεί θα επαληθεύουμε αν η ίδια εκμετάλλευση έχει τουλάχιστον τρεις γεωρικές καλλιέργειες και έχουμε και κάποιες περιόδους οικολογικού ενδιαφέροντος. Πιστεύω μετά θα μπορούμε με, να τις ελέγχουμε πιο καλά. Αλλά αν θέλουμε να είναι πιο μεγάλη ευελιξία κατόπιν αιτήματο κάποιων κρατών μελών, ε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή ε, τομή και μεγαλύτερη ευελιξία και άποψη χωρί. Ε, δηλαδή χωρί πιο μεγάλη πολυπλοκότητα. Θέλουμε να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Θέλουμε να έχουμε και κάποια μέτρα περιβαλλοντικά στον δεύτερο πυλώνα, για παράδειγμα. Μπορεί αυτό να διευκολύνει την κατάσταση. Αν έχουμε έναν γεωργό που έχει κάποια γεωργό περιβαλλοντικά μέτρα, θα μπορεί αυτά να τα ισοσταθμίσει με τα εξισώσει με έτοιμα green, πρασινίσματο. Να μην κάνει δύο φορέ το, ίδιο πράγμα. Βέβαια, το γραφειοκρατικό άχθο θα, θα επηρεαστεί και από το βαθμό ευελιξία που θα ζητήσουν τα κράτη-μέλη για τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου και την πολυπλοκότητα των κανόνων στα κρατη Το έχω πει και πριν. Για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο θα δώσω μεγαλύτερη προσοχή στη δυνατότητα ελέγχου, επαλήθευσης ε, των ε, μέτρων αυτών. Ήδη ξεκινάμε να προβάλλουμε τις καλές και τις κακές πρακτικές για να δούμε πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει απλά το ίδιο μέτρο. για την ανάκτηση έχουμε μια διακύβανση, αλλά από τότε που ισχύει ο κανόνας 50-50 μειώνονται οι διακυμάνσεις αυτές. Για το 2011, από τότε που εφαρμόζεται λοιπόν ο κανόνας 50-50, τα ποσοστά ανάκτησης είναι υψηλότερα. Για το 2011 που βρισκόμαστε, βρισκόμαστε ήδη στο 44% ανάκτησης για όλη την περίοδο. Από τότε δηλαδή που να ισχύει ο κανόνας αυτός. Από το επόμενο δημοσιονομικό δημοσιονομική περίοδο προτείνουμε τον κανόνα το 100% ακριβώς για να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα κράτη-μέλη αφού είμαστε στη μεικτή κοινή διαχείριση. για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις δασικές εκτάσεις ε, και την οριοθέτησή τους, εκεί έχουμε αρκετά σαφείς θα έλεγα κανόνες. Μπορεί να υπάρχει κάλυψη, ε, να έχουμε δηλαδή ένα μέγιστο αριθμό εκτάριου που καλύπτεται από ε, δάσος στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν σαφείς ορισμοί. Πρόβλημα είναι πώς μετράτε η έκταση. Στην επόμενη μεσονομική περίοδο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν πιο ξεκάθαρο ορισμό για τους σκοτόπους για να μην έχουμε και εδώ κίνδυνο λάθους. Τώρα, έλεγχοι επιτόπου. Οι έλεγχοι γίνονται από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν ελέγχει τους ελέγχους, αν θέλετε, των κρατών μελών. Και πού μπορούμε να παρέμβουμε, στην ποιότητα των ελέγχων. Κυρίω ό,τι αφορά το προπαρασκευαστικό έργο που μπορούμε να φέρουμε σε πέρα από κοινού με τα κράτη-μέλη. Για την ανάπτυξη τη Πέθρου τώρα, αναλύουμε το ενδεχόμενο να μπορούμε να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί με όσα κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη του όλε τι συστάσει τη Κομισιόν για να βελτιώσουν του ελέγχου του. Τα στοιχεία αυτά θα τα εξηγήσω στο σχέδιο δράση που θα σα ε, προτείνουμε από εδώ μέχρι την ψηφοφορία για την απαλλαγή. Και υπάρχει επομένω μια ευθύνη, κύριε Μιλντερ, πολιτικού χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη. Εγώ θα έλεγα ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της τελευταίας χρονικής περίοδου, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια διακύμανση στο ποσοστό των σφαλμάτων, αλλά για τον πρώτο πυλώνα μπορούμε να μιλήσουμε για μια σταθεροποίηση μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Από τη στιγμή που εφαρμόστηκε το σύστημα EAS, Ajax, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση σε σχέση με το ποσοστό των σφαλμάτων, γιατί έχουμε και πιο αξιόπιστα δεδομένα. Εκεί που παραμένει κάποιο έργο να φέρουμε σε πέρας είναι ο τομέας της αγροτικής ανάπτυξης, όπου το σύστημα Άγιαξ έχει τα όρια του, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ζητήματα και θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να θεσπίσουμε ένα σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης και μάλλον ε, πιστοποίησης του συστήματος πιστοποίησης έχουμε εστιάσει πολύ την ε, προσοχή μας στον ε, Άγιαξ και λιγότερο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την ε, αγροτική ανάπτυξη, όπου είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος της αποκοινού διαχείρισης από ότι στον τομέα των πληρωμών. Για τις επιχειρήσεις κρατικού χαρακτήρα και τις επιδοτήσεις του, τους, έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις μέσα στο σύστημα μεταρρύθμισης. Ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί, αλλά δεν είναι η έλλειψη θέλησης της Κομισιόν αλλά εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια, μια συνολική συμβαστική λύση. Έχει και το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει κάποιο ρόλο και ελπίζω ότι θα μπορέσει και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να εκφράσει την αποψή τη ενώπιον τη Ολομέλεια για το περιεχόμενο αυτών των ε, προτάσεων. Αυτό Νομίζω ότι απήντησα στο ερώτημά σα. Γιατί είπα ότι το γεγονό ότι έχουμε ένα ποσοστό σφαλμάτων υψηλό σε ορισμένε ε, ε, διαδικασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τα χρήματα. Υπάρχουν ενδεχομένω φάλματα στη διαδικασία, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ανακτηθούν τα χρήματα αυτά. Και αυτά λοιπόν για τις ανακτήσεις, όπως ανέφερα προηγουμένως, στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης θα πρέπει να επομιστούν και τα κράτη-μέλη την, ε, τις ευθύνες τους, γιατί πρόκειται και για χρήματα φορολογουμένων, είτε εθνικών, είτε Ευρωπαϊκο, Ευρωπαίων. Και σε εσά κύριε Οντή, νομίζω ότι απήντησα για την διαφορά μεθοδολογίας μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου και της ε, Κομισιόν για την καταμέτρηση των σφαλμάτων. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση μεθοδολογίας το 2011 και το 2012 και αυτό θα μας δώσει μια σαφέστερη εικόνα γιατί στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης έχουμε μια διαφορά που έχει να κάνει με τον κυκλικό χαρακτήρα των ε, προγραμμάτων ανάπτυξης και είναι πιο έντονη από ό,τι στον πρώτο πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα έχουμε ένα πολυετές επίπεδο σχεδιασμού και τώρα βρισκόμαστε στο επίπεδο κορύφωσης εφαρμογής ορισμένων προγραμμάτων και επομένως αυξάνονται και οι κίνδυνοι στον τομέα αυτό. Και για τον κύριο Όσλιγκ επίσης νομίζω ότι απήντησα. Και για τις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις αλπικού χαρακτήρα εκτάσεις και για τα μέτρα <clears throat> περιβαλλοντικού χαρακτήρα πιστεύω και εγώ ότι μπορούμε να απλοποιήσουμε την εφαρμογή αλλά και τον χαρακτήρα αυτών των μέτρων με το να χρησιμοποιούμε κριτήρια επιλεξιμότητας και να υπάρχει και η δέσμευση από την πλευρά των γεωργών ότι θα εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μειώσουμε τον ποσοστό σφαλμάτων χωρί να υπονομεύσουμε την ποιότητα αυτών των περιβαλλοντικών μέτρων. Θέλω να κλείσω εδώ λοιπόν και σα διαβεβαιώ ότι παίρνω πολύ στα σοβαρά τα προβλήματα αυτά τα οποία αναφέρατε για την αγροτική ανάπτυξη και θα επανέλθω με απαντήσεις στα θέματα αυτά, κυρίως σε ό,τι αφορά για την μεσοπρόθεσμη προοπτική μας και φυσικά θέλω με ενόψη της νέας περίοδου προγραμματισμού να έχουμε βελτιώσεις αλλά ξέρετε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνονται από τον ένα χρόνο στον άλλο. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μια θετική ανέλυξη για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις σας που είναι τόσο σημαντικές για την εργασία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε, επειδή υπήρξε και μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων, έχουμε φτάσει και στα όρια του, του χρόνου μας. Θα πρέπει να κλείσουμε εδώ. Βέβαια αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον των συναδέλφων της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για τα θέματα ελέγχου του προϋπολογισμού αγροτικών θεμάτων, που είναι και το μεγαλύτερο τμήμα του αγροτικού του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ετέθηκε ένα ερώτημα προς το ελεκτικό συνέδριο και δεν ξέρω αν θα μπορούσε το ελεκτικό συνέδριο να μας δώσει μια έγγραφη απάντηση και να εστιάσετε στα κυριότερα θέματα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς, τον, ε, προς την ακρόαση του κυρίου Έτιγκερ. Θέλετε να πείτε κάτι από το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Άγκουστιν. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα ερωτήματα και βλέπω με τα χαράς ότι Έχετε λάβει την έκθεση. Ο κύριο ε, Τσιόλο απάντησε τα περισσότερα ερωτήματα σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη τη μεθοδολογία μας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η περιγραφή της μεθοδολογίας μας είναι στο κεφάλαιο 1 τη έκθεσή μα. Οπότε το καλύτερο που έχω να σας προτείνω είναι να διαβάσετε το κεφάλαιο αυτό. Κεφάλαιο 1. σε ό,τι αφορά την ε, τάση των ποσοστών σφαλμάτων, το ερώτημα πόσο πρέπει να περιμένουμε, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε για τα σωστά δεδομένα. Μα πάντα είναι σωστά τα δεδομένα με βάση τη μεθοδολογία μας. Είναι, αλλά όπως σας είπα, για πρώτη φορά έχουμε μια ξεχωριστή αξιολόγηση για το πρώτο και το, για το δεύτερο πυλώνα. Έχουμε λοιπόν κάνει έναν έλεγχο σε ένα πλήρες δείγμα πράξεων, συναλλαγών. Είμαι σχεδόν βέβαιος λοιπόν ότι τα αποτελέσματα τη επόμενη χρονιά ε, θα παρουσιάζουν μια πραγματική τάση. Αυτά είχα να πω από πλευρά μου. Σας ευχαριστώ. Yeah, ε, for... Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Θα ήθελα να δώσω και σε εσάς κυρία μου το λόγο για ένα σύντομο σχόλιο. Σας ευχαριστώ. Τίποτα δεν έχω να πω στην ουσία σε σχέση και να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Επίτροπος Τσόλος. Θέλω να πω μονάχα για τα θέματα των δεσμεύσεων σε σχέση με το περιβάλλον όπου οι δικαιούχοι δεν εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Δεν κρατούν ζώνες ε, ενδιάμεσες οι οποίες θα είναι ελεύθερες από εμφυτεύσεις. Χρησιμοποιούν λοιπάσματα και κάνουν πολλές άλλες, πολλές άλλες παραδιάσεις των ε, απαιτήσεων που θέτουν τα κράτη-μέλη για την επιδότηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά τη διάρκεια της παρούσης και της ε, επερχόμενης ε, περίοδου. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο, διότι στην ε, έκθεσή σας αναφερθήκατε και στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που αναφέρθηκε και στη συζήτηση, γιατί είναι φανερό ότι με ένα απλούστερο σύστημα θα μειωθεί και το ποσοστό σφαλμάτων και επομένως και η Κομισιόν, αλλά και τα κρατημέλη θα πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομοθέτης επίσης. Έχουμε ήδη κάποιες πολιτικές αιτήσει προς την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι πρόκειται για το θέμα της επιλεξιμότητος, της πολλαπλής συμμόρφωσης, του πρασινίσματος. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία έχουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους και όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι υπάρχουν πολλές μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του αν αξίζει τον κόπο να αντιμετωπίζουν όλη αυτή την πολυπλοκότητα και αν με ένα πλούστερο σύστημα δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Τσόλος. Θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας στην Επιτροπή της, ε, του Ελέγχου του Προϋπολογισμού να είναι προδραστική η Επιτροπή και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τα προβλήματα αυτά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για το γεγονός ότι ήσασταν παρόν σήμερα και ως Άγιος Βασίλης, Άγιος Νικόλαος για το δυτικό σύστημα. Έχετε δώσει πραγματικά ένα σημαντικό δώρο προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έδωσε χρυσά νομίσματα σύμφωνα με τον θρύλο ο Άγιος Νικόλας, εδώ δεν θέλουμε ακριβώς κάτι τέτοιο, αλλά θέλουμε να βοηθήσετε τους γεωργούς στο να μπορέσουν να συνεχίσουν την εργασία τους και να έχουν τη δυνατότητα παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τους. Ε, σε μια εποχή ισχνών αγελάδων βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει και πρέπουσα προσοχή για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα, τα δημόσια κονδύλια. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο. Το κύριο Γκάιερ θέλει να λάβει το λόγο. Θέλουμε λοιπόν να σα ευχαριστήσουμε τα μάλα, κύριε Επίτροπε Τσόλο. Ja, dann darf ich gleich äh, weitermachen mit... Äh, Καλώς. Συνεχίζουμε με τον Επίτροπο Oettinger τώρα. Κύριε Οντή. Oui, Monsieur le Président. Herr Odi hat das Wort. Oui. Έχετε το λόγο, κύριε Οντή. Κοιτάξτε, κανονικά στις 11 ξεκινάμε ψηφοφορίες και προβλέπουμε, ε, ξέρετε, τις, το χρόνο εργασίας μας και το χρόνο ταξιδίου ε, σε σχέση με τα ωράρια τα οποία μας προτείνετε. Γι' αυτό παρακαλώ να σεβαστούμε τον χρόνο που προβλέπετε. Um, vote uh, from 11... Κοιτάξτε, θέλαμε να ψηφίσουμε από τις 11 μέχρι τις 12 και μισή. Είστε όλοι έτοιμοι να ψηφίσετε? Θέλετε να ψηφίσουμε πρώτα? Έχουμε τον κύριο Έτιγκερ εδώ, δηλαδή... Πού πήγε ο Επίτροπος? Καλά, ας ψηφίσουμε πρώτα λοιπόν. Okay, can we vote? Can we vote? If nobody, if yeah, yeah, nobody objects. No? No. Ja, Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στις ε, ψηφοφορίες. Έχουμε καταρχήν την ε, ειδική έκθεση Calfin. Ξεκινάμε. Έχουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 πρώτα. Συμβαστική τροπολογία επαριθμών 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110 με προφορική τροποποίηση. Παρακαλώ. Κύριε Καλφίν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω κάτι στα πλαίσια της ψηφοφορίας. Κάποιες τροπολογίες δεν συνδέονται με τη συγκεκριμένη παράγραφο. Καλό θα ήταν να ψηφίσουμε πρώτα τις συμβιβαστικές τροπολογίες, εφόσον συμφωνούν και οι συνάδελφοι βέβαια, και μετά όλες τις υπόλοιπες. Äh, äh, Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, μπορώ να το κάνω. Είναι δυνατόν. Ε, εντάξει. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία υπαρθμών 4. Ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε την 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Amendment number 21. 21 με 23 Ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 30. Έχει καταπέσει. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 και 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτέ. 39 τώρα υπέρ κατά αποχές δεκτή Σαράντα υπέρ κατά α όχι έχει καταπέσει η σαράντα... έχετε δίκιο Σαράντα τρία... υπέρ κατά αποχές δεκτή τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 46 έχει καταπέσει. Συνεχίζουμε τώρα. Με την 49 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, 49. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55 και 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτής. Συνεχίζουμε με την 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 με προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 και 65 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ε, ξέχασα την 63. Λοιπόν, πηγαίνω πίσω στην 63 και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεχίζω με την 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 117 με προφορική τροπολογία υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 και 82 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτή 84 σε δύο τμήματα και είναι υπέρ του πρώτου τμήματος υπέρ κατά δεκτό το πρώτο τμήμα δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 85 καταπίπτει εφόσον γίνεται δεκτή το 84 86-87 υπέρ κατά, αποχές, δεκτές. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 και 90 υπέρ, κατά. Α, έχουμε ε, προφορική τροπολογία σε τι. Στην 90. Μπορείτε να διαβάσετε παρακαλώ με το μικρόφωνο. Αντί να πούμε στο πλαίσιο, να πούμε επί τη βάση του κανονισμού του 2006. Θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στο πλαίσιο αλλά και στο συγκεκριμένο κανονισμό. Καλώς ε, είδαμε λοιπόν την ψηφίζουμε λοιπόν για την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται η προφορική. Ψηφίζουμε το αρχικό 89 και 90. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 91 και 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Η 95 έχει καταπέσει. Η 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άφετ λοιπόν 1 με 5 μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού. Όχι. Την 1 και 2 λοιπόν της Άφετ υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4 και 5 από κοινού. Α, όχι, μόνο 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος επί της ΑΦΕΤ 5. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ΑΦΕΤ 5. Πέρα της ψηφοφορίας. Καλώς. Δεκτή. Λοιπόν, στον προϋπολογισμό μπορούμε από την 3 μέχρι την 6 να ψηφίσουμε από κοινού. Όχι. Ξεκινάμε λοιπόν με την 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με την 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 και 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 14, όχι, έχει καταπέσει 14. 109 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Όχι, απορρίπτεται. Απορρίπτεται 109. Λοιπόν, η πρώτη αναφορά προϋπολογισμός 1. Κατά. Δεκτή. Τώρα το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Καλφίν. Σας ευχαριστούμε κύριε Καλφίν. Το επόμενο τώρα. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τώρα περνάμε στην έκθεση ΣΤΑΣ. Περνάμε αμέσω στην ψηφοφορία. Παράγραφο 5 ε, στην τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχέ. Ηλεκτρονικό έλεγχο, τροπολογία 1, άρχεται ψηφοφορία. Έχετε ψηφίσει όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ψηφι υπέρ. Κατά, αποχές,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 Ωραία, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη βοήθεια, που ήταν όλοι συγκεντρωμένοι. Και τώρα... Sorry for that. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε αποφασίσει μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ε, απαλλαγής για τον προϋπολογισμό της Κομισιόν του 2011 να προβούμε και σε μια ακρόαση του Επιτρόπου Γκίντερ Έτιγκερ στην Επιτροπή μας. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας καλωσορίσω εξ ονόματος της Επιτροπής μας για το ελεκτικό συνέδριο είναι ο κύριος Αρικέτεν, ο οποίος θα είναι πάρον επίσης. και θα ήθελα όπως ε, είναι τα Ιωθώτα να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Γκάιερ ως εισηγητή για την απαλλαγή του 2011. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έτιγκερ για την παρουσία του σήμερα το πρωί. Ζητούμε συγγνώμη γιατί κάπως μπερδεύτηκε το χρονοδιάγραμμά μας σήμερα γιατί οι συζητήσεις που είχαμε με τον ε, συνάδελφό σας, τον κύριο Τσόλος, ίσως κάπως ε, τράβηξαν λίγο περισσότερο και ήταν πιο πολύπλοκες γιατί ίσως είναι πιο μεγάλες οι ανησυχίες μας στον αγροτικό τομέα από ό,τι στον τομέα της ενέργειας. Δεν θέλω τώρα να κάνω εισαγωγικές παρατηρήσεις. Απλώς να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή που μου έδωσε ο πρόεδρος στον λόγο να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Να, να τη χρησιμοποιήσω για να θέσω ερωτήματα. Στο παρελθόν η Επιτροπή μας έχει αντιμετωπίσει δύο ζητήματα που εμπλέκονται στο δικό σας τομέα αρποδιοτήτων. Πρώτον, η εξέλιξη του κόστους για το πρόγραμμα ITER, e για την πυρηνική σύνδεξη, γενικότερα για την ε, πρόθεση των παγκοσμίων σχεδίων για την πυρηνική σύνδεξη. Το ITER e είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο λοιπόν στα ερευνητικά προγράμματα αυτού του είδους και δεύτερον είναι οι εξελίξεις για την θέση σε αχρηστία πυρηνικών σταθμών στη Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία των πυρηνικών σταθμών που είναι του ίδιου τύπου με τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ. Ένα τρίτο ερώτημα είναι η αύξηση των σφαλμάτων που παρατηρούνται στην εκτέλεση της πολιτικής έρευνας. Έχουμε ήδη ακούσει από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου και εμείς προσπαθήσαμε κάπως να καταμερίσουμε αυτά τα προβλήματα με τη βάση του ποια υπηρεσία της Κομισιόν ασχολείται με τα θέματα αυτά. Βλέπουμε ότι στη Γενική Διεύθυνση Ενεργείας ότι υπάρχει αύξηση και του ποσοστού σφαλμάτων κατά που έχει φτάσει στο 4,5% και θα θέλαμε για αυτό το λόγο να συζητήσουμε μαζί σα για να ξέρουμε ποιε είναι οι σκέψει από την πλευρά τη Κομισιόν για το πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί ο αριθμό αυτό των σφαλμάτων και επίση θα θέλαμε να ξέρουμε από τη δική σα πλευρά ποια είναι τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε ένα υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων στην ενεργειακή πολιτική από ό,τι σε άλλου τομεί πολιτική. Επανέρχομαι και πάλι στη θέση αχρηστία πυρηνικών σταθμών. Η Επιτροπή μα έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό πολλές φορές πήγε και στην Ιγναλίνα στη Λιθουανία, σχεδιάζει στα, στις αποστολές μας του χρόνου να επισκεφθεί τους άλλους πυρηνικούς σταθμού στην Βουλγαρία και στην Σλοβακία που πρέπει να τεθούν σε αχρηστία. Στην Λιθουανία είχαμε κάπως το αντίστροφο πρόβλημα από ό,τι πολλές άλλες φορές. στην περίπτωση της Λιθουανίας δεν είναι ότι δόθηκαν τα χρήματα με λαθασμένο τρόπο, απλώς δεν δόθηκαν καθόλου. Εμάς δεν μας ικανοποιεί γιατί με τον τρόπο αυτό δεν επετεύχθη ο στόχος που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, ήθελα να ξέρουμε, θα να ξέρουμε ποια είναι η εκτίμηση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μεταξύ Λιθουανίας και των συμβατικών της εταίρων. Για το ίτερ επίσης μπορεί να θέσει κανεί το μεθοδολογικό ερώτημα του αν τίθεται σε κίνδυνο η ενότηση του προπολογισμού εφόσον το ίτερ παραμένει και πάλι <clears throat> εκτός του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εγώ θέλω να θέσω και ένα περαιτέρω ερώτημα. Θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η αύξηση του κόστους του ίτερ είναι ελεγχόμενη. Γιατί τα κράτη-μέλη βλέπουν να έχουν την τάση την αύξηση του κόστους του ΙΤΕΡ να την καταλογίζουν στο συνολικό προϋπολογισμό έρευνας. Και αυτό δεν τους οδηγεί σε κανένα, καμιά προσπάθεια να αντιμετωπίσουν περισσότερο προσεκτικά την ε, έρευνα στον τομέα αυτό και δεν θέλουν να περιστήλουν το κόστος του ΙΤΕΡ. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω στον Αρή Γκρετέν το λόγο. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε επειδή ο εισηγητή σα έχει ήδη θέσει ερωτήματα που ήθελα να θέσω και εγώ ίδιος, για να συντομεύσω τη συζήτηση θα απαρνηθώ της ανάγκης να θέσω ερωτήματα. Έχω τον γραπτό λόγο μου στη διάθεσή σας εάν θέλετε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Βλέπω ότι το ελεκτικό συνέδριο προχωρεί σε εξοικονομήσεις ήδη. Οπότε μπορώ να δώσω κατευθείαν το λόγο στον Επίτροπο κύριο Έτιγκερ και να τον παρακαλέσουμε να απαντήσει και στα ερωτήματα που έθεσε ο εισηγητής μας. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκάιερ, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, κύριε Γκρέτρεν και εκπρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν να σας τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας από ιστορική άποψη ήταν μια πορεία προς τη ρύθμιση, προς την θέσπιση στόχων, απαγορεύσεις και αδειοδοτήσει. τώρα τα τελευταία χρόνια αποκτά ένα ιδιαίτερο ρόλο και μέσα στην πολιτική ε, προϋπολογισμού. Αναφέρθηκε ήδη το πρόβλημα, το πρόγραμμα Ίτερ, υπάρχουν μεγάλα σχέδια λοιπόν όπως το Ίτερ και η πρόταση τη Κομισιόν για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, τα επόμενα 7 χρόνια, έχει τρία κύρια σημεία εστίασης την ε, σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού και τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο λοιπόν. Είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της χρήσης ενέργειας, η εξυγίανση των κτίριων, όπου θα υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία του προϋπολογισμού, υπάρχει διευκόλυνση Connecting Europe, δηλαδή η πρόταση της Κομισιόν για τη βελτίωση των υποδομών ενέργειας και διασύνδεσης για να υπάρξει μια καλύτερη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου και των υποδομών και επίσης θέλουμε να παροτρύνουμε μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα της ενέργειας. Θέλω να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για την ετήσια έκθεσή του και την ανάλυση που μας έχει παρουσιάσει και επίσης για την ειδική έκθεση σε ό,τι αφορά την θέση σε αχρηστία πυρηνικών σταθμών. Έχουμε το θέμα αυτό των πυρηνικών σταθμών σε τρία κράτη-μέλη που θεσπίστηκε ως στόχος ήδη από την είσοδο των χωρών αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να υπάρξει μια συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αυξηθεί και το επίπεδο ασφαλείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Χρησιμοποιούμε την ε, εμπειρογνωμοσύνη και τη βοήθεια της ε, τράπεζας αυτής για να επιτύχουμε το στόχο αυτό της θέσης σε αχρηστία των στόχων. Υπάρχουν τώρα 13 συγκεκριμένα μέτρα που καλύπτουν περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία τίθενται προς την κατεύθυνση αυτή σε χρησιμοποίηση στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία. 50% των μέσων αυτών έχουν εφαρμοστεί, στη Λιθουανία μόνο το 30%. Εδώ ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της προσπάθειάς μας ήταν όχι μόνο να εξυπηρετήσουμε την διαδικασία αχρήστευσης και διάλυσης αυτών των σταθμών, αλλά συγχρόνως να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια εφοδιασμού με ενέργεια, την αποδοτικότητα των ε, διάφορων θερμικών σταθμών, δημιουργία ενός νέου σταθμού που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο στη Λιθουανία. Από τη μία πλευρά λοιπόν θέλουμε να αφαιρέσουμε από την λειτουργία τον πυρηνικό αντιδραστήρα, από την άλλη μεριά να υποστηρίξουμε την υποδομή παροχής ενέργειας και ηλεκτροδότησης, ώστε να εξασφαλίσουμε για τους πολίτες την ασφάλεια εφοδιασμού με ενέργεια. Για τα θέματα θέση σε αχρηστία, τα προπαρασκευαστικά μέτρα έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους και έχουν σχεδιαστεί και οι σταθμοί υποδοχής των αποβλήτων. Έχουν προχωρήσει λοιπόν οι ενέργειες για την εκένωση αυτών των σταθμών και έχουν ξεκινήσει και οι προσπάθειε για την μετασκευή του. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι ότι κατά την άποψή του προχωρά με βραδύ ρυθμό η διαδικασία αυτή θέση σε αχρηστία. Εμεί είμαστε πάντα σε επαφή με τι αρχέ τη Λιθουανίας σε επίπεδο υπουργών και σε επίπεδο τεχνικό. Και η εντύπωσή μα είναι ότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση τη Λιθούανία να φέρει σε πέρα στις συμβατικέ τη υποχρεώσεις. και δεν υπάρχει καμία τακτική καθυστέρησης και βραδιπορίας, ούτε μια προσπάθεια να τεθεί και πάλι σε εφαρμογή, να χρησιμοποιείται και πάλι ο πυρηνικός σταθμός. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η δυσκολία που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Ενέργειας Λιθουανίας λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις οι οποίες συνδέονται με τη θέση αγριστία του σταθμού αυτού. Επομένως μας έχει προσκαλέσει Μα προσκάλεσε να παίξουμε και κάποιο ρόλο στο Υπουργείο στο Εθνικό Υπουργείο Ενέργεια τη Λιθουανία. Εμεί βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να παραμείνουμε σε επίπεδο ουδετερότητα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Τώρα η νέα κυβέρνηση έχει προβλέψει να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνιστεί και εμείς επομένως θα αναμείνουμε να υπάρξει και μια κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης της Λιθουανίας. Φυσικά υπάρχει μια πολιτική πίεση από ορισμένου να τεθεί και πάλι σε, σε λειτουργία ο πυρηνικός αυτός σταθμός μετά από την κρίση εφοδιασμού σε φυσικό αέριο με το 2009. Αλλά όλες οι κυβερνήσεις έχουν απόλυτη επίγνωση της ανάγκης ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της θέσης σε αγριστία αυτού του πυρηνικού σταθμού το αργότερο του χρόνου. Από την πλευρά του ελεκτικού συνεδρίου Εμείς δεχόμαστε όλα αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί εκεί και θεωρούμε ότι όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη πλήρως στην εργασία μας. Υπάρχει ένα σημείο βέβαια το οποίο ενδιαφέρει και το Κοινοβούλιο. Υπάρχει πρόβλεψη περαιτέρω κονδυλίων στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα τρία αυτά κράτη-μέλη για τη θέση αριστεία των ποινικών σταθμών που θεωρούνται και από τις τρεις εμπλεκόμενες χώρες ως ιδιαίτερα χαμηλά αυτά τα ποσά. Επίσης παραμένει ανοιχτό το θέμα του αν θα πρέπει να συνεχίσει η χρηματοδότηση με τις μελλοντικέ πολιετές, πολιετής ε, προοπτικές, αν θα είναι η επόμενη περίοδος η τελευταία ή αν και επέκεινα του 2020 θα μπορέσει να υπάρξει χρηματοδότηση αυτού του είδους. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πίεση ώστε να σταματήσει η χρηματοδότηση με, τις επόμενες, ε, με την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. ΉΤερ. Το Ίτερ είναι ένα μοναδικού χαρακτήρα εγχείρημα και από το οποίο πρέπει να αποκομίσουμε και εμπειρίες. Η Κομισιόν παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία αυτή. Η σύνδεξη για την ενέργεια είναι ένα από τα βασικά μας σχέδια όπου εμπλέκονται μεγάλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία. Έχουμε επίσης έξι μεγάλους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ιαπωνία, Κορέα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα, Ρωσία, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό το ITER. Και ο Γενικός Γραμματέας για τα θέματα αυτά, όπως και εγώ ο ίδιος έχουμε έλθει σε επαφή με όλους αυτούς τους εταίρους για να προχωρήσουμε τη συνεργασία μαζί του συμμετέχουμε σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου για τα θέματα αυτά. Έχουμε ένα νέο διευθυντή τώρα για τα θέματα του προγράμματος Fusion for Energy, ο οποίος ε, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Και μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, είναι στη διάθεσή σας να έλθει να σας παρουσιάσει τα θέματα αυτά. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει πολύ υψηλή διαχειριστική ικανότητα. Και έχουμε φυσικά πάρα πολλούς επιστήμονες υψηλού επίπεδου στο πρόγραμμα ITER. Το θέμα όμως της διαχείρισης, το θέμα της περιστολής του προϋπολογισμού δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς μέχρι στιγμής και ελπίζω ότι αυτός ο νέος διευθυντής του Fusion for Energy θα μπορέσει να αναπτύξει περισσότερο τις ε, ικανότητες διαχείρισης στο ITER και να οδηγήσει και σε μεγαλύτερη επίγνωση των προβλημάτων του προϋπολογισμού για τα θέματα της ε, ενέργειας και ότι θα μπορέσει το νέος αυτός διευθυντής να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του πλήρως. Ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε μέσα στα πλαίσια των στόχων του προϋπολογισμού. Η πρόταση της χρηματοδότησης του ΙΤΕΡ μέσα στον προϋπολογισμό ήταν η θέση της Κομισιόν. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε ότι η χρηματοδότηση αυτή έχει επιβληθεί μέσα στον προϋπολογισμό έρευνας από τα κράτη-μέλη. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι οποιοδήποτε ευρώ το οποίο βρίσκεται μέσα στον προϋπολογισμό του ιτερ σημαίνει περικοπή των άλλων μορφών έρευνας εκτός του ιτερ και επομένως θα πρέπει να μην βρίσκονται τα προγράμματα ενέργειάς μας πάντα υπό τη δεμόκλειο σπάθη της αύξησης των κονδυλίων του ΙΤΕΡ. Εγώ λοιπόν έχω κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσω μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ανάγκης να προχωρήσει το σχέδιο αυτό, αλλά με ελεγχόμενη χρηματοδότηση και όχι σε βάρος άλλων ε, μορφών χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων ενέργειας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Επίτροπο. Θα ήθελα τώρα να δω αν θα ήθελε κάποιος να θέσει ερωτήματα προς τον κύριο Επίτροπο. Προς το παρόν δεν βλέπω κάποιος να θέλει να θέσει ερωτήματα. Ναι, ο κύριος Κάλφιν μονάχα θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πράγμα να ρωτήσω τον κύριο Έτιγκερ. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα θέμα εδώ πολιτικής βούλησης, γιατί σε ορισμένες χώρες τα τεχνικά προγράμματα προχωρούν πέραν του 2020. Όταν λέτε ότι αυτά θα πρέπει να τελειώσουν μέχρι το τέλος του 2020, αυτό είναι θα έλεγα συμβατό με τις τεχνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια. Uh, Ευχαριστώ κύριε Κάλφιν. Και εγώ είχα θέσει αυτό το ερώτημα όταν είχαμε πάει με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στη Λιθουανία και μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι ότι εμείς ως ε, εκπρόσωποι της Επιτροπής Προϋπολογισμών πήγαμε στην Ιγναλίνα και θέσαμε πολλά ερωτήματα γιατί η εντύπωσή μας ήταν ότι ε, υπήρχε κάποια προσπάθεια να ρυφθεί αλλού το βάρος της έλλειψης πρόοδου για τα θέματα αυτά. Είσαστε λοιπόν έτοιμος να αλλάξετε τις δομές διαχείρισης που θα εξασφαλίσει ότι θα γίνει εγκαίρος μέχρι το 2020, δηλαδή η θέση στην ε, συναχρηστία αυτού του πυρηνικού σταθμού και είχαμε την εντύπωση ότι χρειάζεται και κάποια διαδικασία διαμεσολάβησης ώστε να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν σε ένα κοινό σχέδιο. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα του ταξιδίου μας στην Ιγναλία και εδώ και η κυρία Χέρτσοκ να, να λάβει το λόγο σχετικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το ίδιο θέμα Θέλω και εγώ να κάνω ένα ερώτημα, διότι μάθαμε στη Λιθουανία και για κάποιου ε, τρίτου εταίρου, συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την, για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, την BERD, ως ε, εταίρο. Άρα έχουμε συνεργασία με την Εθνική Κυβέρνηση κτλ. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και έχω και ένα ακόμη ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά την ε, Ευρώπη βρισκόμαστε λίγο πίσω σε ό,τι αφορά και τον παροπλισμό τέτοιων εγκαταστάσεων. Ε, εξού και οι καθυστερήσεις αυτές. Διότι είναι λιματικός ο κλάδος, αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λοιπόν, και από οικονομικής πλευράς ε, να τα βγάλουμε πέρα με την ε, αιτήσια διαδικασία κατάρτισης προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το project αυτό. Πώς ε, θα θέσουμε σε χρηστή αυτό το σταθμό με απόλυτη ασφάλεια τους πολίτες, γιατί αυτό είναι από το στόχος. Ja, äh, Δεν βλέπω να θέλει κανείς να λάβει το λόγο περαιτέρω. Μπορώ να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Πίτροπο να μας παρουσιάσει απόψη του για το θέμα αυτό. η δομή της συνεργασίας σε σχέση με τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ε, πλοκή. πολύπλοκη. Εγώ είχα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στην, ε, ε, να επιφορτήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση και με τη διαχείριση της διαδικασίας αυτής. Βέβαια, η Λιθουανία πρέπει και αυτή να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και είναι φανερό ότι δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή ένα τόσο μεγάλο σχέδιο να το εφαρμόσει επαρκώς σε καθημερινό επίπεδο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα μόνοι μας να φέρουμε σε πέρα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς την συμμετοχή της Λιθουανίας. Οι πληρωμές τώρα και οι καθυστερήσεις που αφορούν το θέμα αυτό Μπορούμε να περικόψουμε ή να ακυρώσουμε τις καταβολές χρηματοδότηση προς τη Λιθουανία, αλλά αυτή τη στιγμή τα οικονομικά αυτά μέσα είναι κατά κάποιο τρόπο το μεγαλύτερο κίνητρο που έχει η Λιθουανία να φέρει σε πέρας αυτό το σχέδιο. Υπήρξαν και διαμάχες μεταξύ της κυβέρνησης και των τεχνικών ομίλων που είχαν αναλάβει τη διαδικασία αυτή και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Χέρτσοκ για το θέμα αυτό. Είτε έχει είτε δεν έχει πυρηνικού σταθμού μια χώρα, η διαδικασία παροπλισμού ενός πυρηνικού σταθμού είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο εγχείρημα. Στην Γαλλία δημιουργούνται νέοι σταθμοί, αλλά υπάρχουν και παλιότεροι οι οποίοι παροπλίζονται. Επομένως, η κατασκευαστική βιομηχανία και η βιομηχανία του, πυρηνικ... του πυρηνικού τομέα θα πρέπει να παραμένουν σε επαφή για να διατηρήσουμε τις απαραίτητες ικανότητες και τις μεγάλες μονάδες οι οποίες είναι σε θέση να αναλάβουν μια τέτοια μεγάλη πρόκληση όπως είναι η θέση ε, αχρηστία ο παροπλισμός πυρηνικών σταθμών. Εταιρείες όπως η Αρέβα, παραδείγματος χάρη, έχουν κάθε συμφέρον να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το έργο του παροπλισμού πυρηνικών σταθμών και όχι απλώς την κατασκευή νέων σταθμών. Αλλά σε εταιρείες όπως η Πίλφιγκερ, επίσης. Το επόμενο χρόνο έχω την πρόθεση να δημιουργήσω μια στρογγυλή τράπεζα σε σχέση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να τους μιλήσω για τα θέματα της έρευνας και της δημιουργίας τεχνικών ικανοτήτων, αλλά επιπλέον και για τα προγράμματα χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ανάπτυξη στο βιομηχανικό τομέα και αυτό αφορά και τη δημιουργία αλλά και τον παραπλησμό πυρηνικών εγκαταστάσεων για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στην πυρηνική βιομηχανία στην Ευρώπη και εγώ πιστεύω ότι το 2020 θα πρέπει να είναι μια οριακή ε, ημερομηνία. Βέβαια και επέκεινα του 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει ένας εταίρος για την χρηματοδότηση σχεδίων όπως το ίτερο. Αλλά όταν βλέπει κανείς την επόμενη ε, δεκαετία και μιλάει και πάλι για συγχρηματοδότηση, αυτό δεν ευνοεί την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία σε χώρε όπω η Λιθουανία. Δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να περιμένουμε στο 2020. Η κυρία Γκρέσλε θέλει να θέσει ένα ερώτημα, όχι για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ, λέει κυρία Γκρέσλε. Αναφέρατε μια συνάντηση στις 15, στις 5 Δεκεμβρίου συγχρόνου συγγνώμη, που ήταν χθες από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχουν κάποιες καταληκτικές προθεσμίες και αν πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να βελτιωθούν τα πράγματα αυτά. Εμείς ήμασταν παρόντες στη Λιθουανία Τρίτη, Τετάρτη και την Παρασκευή θα γινόταν μια συνάντηση που περιμέναμε ότι θα οδηγήσει σε κάποιες προόδους. Γι' αυτό θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα για την κατάσταση όσο έχει τώρα και νομίζω ότι η Κομισιόν είναι υπερβολικά υπομονετική. Στην Λιθουανία δεν έχουμε μόνο ένα σταθμό που τον διαχειρίζεται μια εθνική αρχή, αλλά επίσης υπάρχει και μια νέα κατασκευή η οποία δημιουργείται και εμείς την έχουμε κατά κάποιο τρόπο ανεχθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία ε, θα προκύψουν και ξέρουμε ότι και το κόστος της ε, καθυστέρησης φαίνεται ότι είναι της τάξης των 300.000 ευρώ. Επομένως έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το επιλύσουμε. Έχουμε τα δύο θέματα. Τι κάνετε με αυτές τις νέες κατασκευές και το δεύτερο ερώτημα είναι οι τελευταίες αυτές προσπάθειες να υπάρξει κάποια λύση για το θέμα αυτό, αν πράγματι καρποφόρησαν και αν έχουν προωθήσει τα πράγματα. Και η κυρία Χέρτσοκ και πάλι θέλει να λάβει το λόγο. Πολύ σύντομα. Εγώ υποστηρίζω αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλε. Από την άλλη πλευρά όμως θέλω να δούμε και το άλλο, την άλλη όψη. Δηλαδή έχουμε ένα γενικό πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη παροπλισμού κάποιων πυρηνικών σταθμών. Δεν υπάρχει όμως τεχνική λύση όριμη. Επομένως πρέπει οι σταθμοί αυτοί να κλείσουν γιατί δεν υπάρχει λύση. Δεν έχει βρεθεί κάποια λύση μέχρι στιγμής. Άρα είναι καθαρά για λόγους ασφαλείας και πρέπει να γίνει. Όμως πώς θα το διαχειριστούμε για να μην ε, υπολογιστεί ως φάλμα, ως ε, παρατυπία, ως καθυστέρηση, δεν ξέρω εγώ. Έχουμε εδώ συγκεκριμένα το εξή θέμα. Κάποιες μεμονωμένες λύσεις ε, είναι συνθήσεις οι οποίες λύσεις ενέχουν μεγάλο βαθμό κινδύνου. Υπάρχουν και ζητήματα διαχείρισης όμως. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και να χρηματοδοτήσουμε διαφορετικά τις προσπάθειες αυτές, διότι καταλήγουμε στο ίδιο θέμα όπως με το ίτερ για παράδειγμα, δηλαδή όλο και πιο μεγάλο είναι το κόστος, αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και δεν μπορούμε να καλύψουμε και το κόστος αυτός με βάση τις δυνατότητες που έχουμε. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλερ και η κυρία Χέρτσοκ. Έχουμε αναφέρθει και στη δυνατότητα να υπάρξει ένα πάγωμα των κονδυλίων ως μέσο πίεσης κατά της Λιθουανίας. Αλλά βέβαια ούτε και αυτό είναι ικανοποιητικό γιατί με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε λύσει το υποκείμενο πρόβλημα, το πρόβλημα της ασφάλειας. Και εάν συνεχίσει η κατασκευή αυτού του κτηρίου και θεωρηθεί ότι δεν έχει κατασκευαστεί βάσει των ε, προδιαγραφών, και αν δεν υπάρχει καμία θέληση από την πλευρά της, ε, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό αυτό να προχωρήσει στον παροπλισμό, εμείς δεν καταλήγουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, επομένως ένα πάγωμα των ε, κονδυλίων ε, θα στρέφεται εναντίον των ενδιαφερομένων μεν, αλλά είναι απαραίτητο να δούμε και η Κομισιόν με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ασκήσει πίεση και αν θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα από τη δική της πλευρά, γιατί από την πλευρά του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι σαφές με την έκθεσή του ότι πρέπει να υπάρξει κάποια δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε εμείς ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση εμπλοκής η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην ε, Λιθουανία, αλλά θα πρέπει φυσικά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο να παίξει ένα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πολύ στενές επαφές για τα θέματα αυτά και φυσικά εμείς θέλουμε και να αναλάβουμε δράση αλλά και να ασκήσουμε πίεση στις λιτουανικές αρχές. Εγώ δεν θέλω να οδηγήσω σε πηχαίους τίτλους εφημερίδες με το να τιμωρήσω μέσα σε εισαγωγικά την κυβέρνηση της Λιθουανίας. Αλλά θέλω σας τονίσω ότι εξακολουθώ να έχω πολύ στενές επαφές με τις αρχές της ε, ε, Λιθουανίας. Θα συνεχίσω και με τη νέα κυβέρνηση, με τη νέα αρμόδια υπουργό. Σήμερα είχαμε συζητήσεις για το αν θα πρέπει να υπάρξουν περικοπές των ε, κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσω να σας πω ποια είναι τα ορίσματα στα οποία καταλήξαμε στη συζήτηση αυτή. Προφανώς όμως εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τέτοιου είδους μέτρα. Κυρία Γκρέσσα και πάλι. και πάλι το θέμα της κατασκευής η οποία γίνεται στον σταθμό αυτό της Ιγναλίνας. Εγώ νομίζω ότι ήδη η συνάντηση τελευταίας ευκαιρίας θα γινόταν ήδη τον Ιούλιο και έχει μεταφερθεί, μεταφέρθηκε σε αυτό το μήνα. Δηλαδή είναι πολλές οι τελευταίες ευκαιρίες που δίνονται στη Λιθουανία. Το γνωρίζει η κυβέρνηση της Λιθουανίας ότι δεν είναι ο φορέας αυτός ο οποίος δημιουργήθηκε η καλύτερη λύση για τη διαχείριση του προβλήματος. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του συμμετέχοντας σε αυτά τα σχέδια ως Κομισιόν. Εμείς μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του επόπτη, μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του Συμβούλου, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στην δομή αυτού του φορέα. Αλλά διατηρούμε μια στενή επαφή με την κυβέρνηση για το πώς θα μπορέσουν να γίνουν οι τροποποιήσει αυτή τη διαχειριστική δομή για τον παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού. Και πρέπει η κυβέρνηση της Λιθουανίας να δημιουργήσει μια ειδική μονάδα, μια μικρή μονάδα με ικανούς συνεργάτες η, οποίες οποία μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση και να τη συμβολεύσει για το πώς θα μπορέσει να γίνει η διαδικασία αυτή παροπλισμού. Πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα άρδιν αυτή τη στιγμή. Αλλά ελπίζω ότι θα κατανοήσετε ότι για ένα μικρό κράτος μέλος θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη υπομονή. Από ένα μεγαλύτερο κράτος μέλος θα μπορούσαμε να είμαστε πιο απαιτητικοί από ό,τι έναντι της Λιθουανίας. Αλλά η Κομισιόν ακόμα επιφυλάσσεται για να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος για το θέμα του παροπλισμού του ποινικού σταθμού στη Λιθουανία. Ο κύριος Γκρέτενος, εκπρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου, θα ήθελε να λάβει το λόγο για τα άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εμείς ως Ελεκτικό Συνέδριο έχουμε εκπονήσει και μια ειδική έκθεση για το θέμα της θέσης αχρηστίας του παροπλισμού του, των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη και ο κύριος Σέτιγκερ ανέφερε ότι η Κομισιόν έχει απόλυτα δεχτεί τις προτάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, ως εκ τούτου δεν έχω να σας προσθέσω τίποτα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα τότε να ευχαριστήσω, πριν, προηγουμένως να ζητήσω από τον εισηγητή αν έχει να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και έχουμε καθυστερήσει, οπότε μπορώ ε, να περιοριστώ στο να μην προσθέσω τίποτα. Κρίμα, κρίμα. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη διαδικασία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Γκίντερ για την παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μας. Η ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα ολοένα πιο σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέργεια και με μεταφορικό τρόπο. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία για τις ενέργειες της και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ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 Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να περάσουμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, στην ειδική έκθεση για τη χρήση διαδοτικών ταμείων και ταμείου συνοχής για τη χρηματοδότηση υποδομών σε θαλάσσιους λιμένες. Πρέπει να το αναβάλουμε αυτό το σημείο απουσία του εισηγητή. Ε, έχουμε όμως τις ε, καταληκτικές ε, προθεσμίες για την ε, θα τις αλλάξουμε τις προθεσμίες για τις τροπολογίες ή όχι. Λοιπόν, η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες θα πρέπει να αναβληθεί και αυτή, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την κατάθεση τροπολογιών. Και έρχομαι τώρα στο σημείο 8. Ανταλλαγή απόψεων με τον επικεφαλής της ΟΛΑΦ είναι ο κύριος Γιωβάνι Κέσλερ, τον οποίο καλωσορίζω εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να γίνετε πιο ορατός με το να έρθετε εδώ στα προεδρικά έδρανα. Ο κύριος Κέσελ μας είχε στείλει μια επίστολη και είχε ζητήσει να μπορέσει να παρουσιάσει τη θέση της ΟΛΑΦ για ορισμένα σημεία που είχαν αγερθεί και ο κύριος Κέσλερ θα αναφερθεί σε ορισμένα ζητήματα που άπτονται της διαθεσμικής συμφωνίας και τον έχω ζητήσει να είναι σύντομος λόγω του, της καθυστέρησης στο χρονοδιάγραμμά μας. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ξέρετε ότι είχατε συναντηθεί με τους συντονιστές σε μια κλειστή συνεδρίαση και είχατε ζητήσει να έχετε τη δυνατότητα σε μια δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας να αναφερθείτε. Και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα αυτή και σας δίνω με μεγάλη χαρά το λόγο. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την δυνατότητα που μου δίνετε να είμαι εδώ σήμερα. Νομίζω ότι είναι χρέος μου, έτσι το αντιλαμβάνομαι ε, πρώτα απ' όλα να έρθω εδώ μετά τις συζητήσεις ε, τις οποίες είχατε και την ακρόαση ε, που είχατε διοργανώσει. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι χρέος μου ως ένδειξη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο, προς την Επιτροπή σας και για να υπάρχει και λογοδοσία του Γενικού Διευθυντού της Όλαφ και προς όλα τα θεσμικά όργανα αλλά και προς το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα και προς διευκρίνηση, ε, δηλαδή θεώρησα ότι πρέπει να, τουλάχιστον να προσπαθήσω και εγώ να συνεισφέρω στο να διευκρινιστούν και να διαλυθούν κάποια σύννεφα που φαίνεται ότι υπάρχουν, κάποιο μίχλι που φαίνεται ότι υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες. Πώς να το πω αλλιώς να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο δηλώσεων, πληροφοριών που δεν είναι πλήρης, είναι μερικές, υπενιγμών, νίξων και τα λοιπά που τελικά καταλήγουν να γράφονται στις εφημερίδες ως ειδήσει. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να αντιληφθείτε και τη δική μου παρέμβαση, ότι δηλαδή θα σας παρουσιάσω κάποια πραγματικά περιστατικά. Αυτό θα είναι πιο εύκολο για μένα και για εσάς σε σχέση με ορισμένα σημεία τα οποία έθιξαν Παραδείγματο χάρη Υποπτική Επιτροπή στην ακρόασή σας πριν από ένα μήνα. Το πιο σοβαρό ίσω θέμα, το πρώτο θέμα που θέλω να σχολιάσω, είναι η πρόσβαση της Επιτροπής, ε, της Επιτροπής στα δεδομένα. Θέλω, επαναλαμβάνω, να σας δώσω στοιχεία. Και μπορώ να σας πω ότι από την 1η Φεβρουαρίου την ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία ξεκίνησε η εσωτερική αναδιοργάνωση της Όλαφ, οπότε και η νέα αποπτική Επιτροπή άρχισε τη δουλειά της. Το Γενάρη θα έλεγα, μάλλον, αλλά τέλος πάντων από το Φεβρουάριο και μέχρι πριν από λίγες ημέρες, λάβαμε από την αποπτική Επιτροπή 49 αιτήματα πρόσβασης σε φακέλους. Ή πληροφορίες για το περιεχόμενο των φακέλων. Όλα τα αιτήματα γίνονται δεκτά. Άρα, οποιοδήποτε φάκελος ζητήθηκε, χορηγήθηκε πρόσβαση για αυτόν, ούτε ένας, για ούτε έναν φάκελο δεν αποκρύψαμε στοιχεία ή δεν εμποδίσαμε την πρόσβαση προς την ε, ελεγκτική εποπτική αυτή επιτροπή. Πλήρης διαφάνεια λοιπόν από τη δική μας πλευρά και αυτό θέλω να το τονίσω. Προβλήματα υπήρξαν. Υπήρξαν προβλήματα κατά το παρελθόν δηλαδή από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι το Σεπτέμβριο και αυτό φιλόταν στο γεγονός ότι μόλις είχε ολοκληρωθεί η εσωτερική αναδιοργάνωση της Όλαφ και η Επιτροπή αυτή ουσιαστικά μόλις είχε αρχίσει να μορφώνει άποψη σε σχέση με τις διαδικασίες και τις μεθόδους. Δεν υπήρχε κάποια διαδικασία. Και γι' αυτό είχαμε και καθυστερήσεις. και σε κάποιες περιπτώσεις η Επιτροπή αυτή εποπτεία ζήτησε πρόσβαση σε κάποιους φακέλους, αλλά επαναλαμβάνω τελικά κανένας φάκελος δεν κρα... Ε, υπήρξε που να μην δοθεί στην ε, Επιτροπή αυτή. Από το Σεπτέμβριο και μετά προβλήματα δεν αντιμετωπίσαμε. Άρα όλα βαίνουν ομαλώς από εδώ και πέρα. Γιατί, γιατί τελικά το Σεπτέμβριο υπήρξε γραπτή συμφωνία μεταξύ ημών και της Επιτροπής Εποπτείας για την πρόσβαση στα δεδομένα. Ο φαινόμενος με τον πρόεδρο Τίμερμαν ήταν κάτι που επεξεργαζόμαστε επί μήνες και τελικά το πετύχαμε. Και έτσι δημιουργείται μια διαδικασία, χρειαζόμαστε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορεί η Επιτροπή Εποπτείας να έρχεται σε... Ε, να μπορεί να μελετά τα στοιχεία με το σωστό τρόπο σεβόμενοι όμως ε, και ε, τις διατάξεις ε, κανονισμού 45-2001. Και είχαμε και την, ε, τις διατάξεις που ορίζονται και από τον Ευρωπαϊκό Αποπτή Δεδομένων, τι οποίε πρέπει να τηρεί η Επιτροπή Εποπτεία όταν έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Βέβαια, αυτή η διαδικασία δεν υπήρχε και η συμφωνία σχετική δεν υπήρχε πριν το Σεπτέμβριο, εξού και καθυστερήσει και κάποιες συζητήσεις που είχαμε με την Επιτροπή Εποπτείας. Τώρα όμως, τώρα όμως δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Από το Σεπτέμβριο και μετά, επαναλαμβάνω, κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω να κάνω μια ιδεολογική συζήτηση αν έχουν δικαίωμα άμεσης πρόσβασης κτλ. κτλ. Είναι κάτι το οποίο μάλιστα ζήτησαν πρόσφατα με επιστολή τους. Αυτό είναι θέμα των θεσμικών οργάνων και συγκεκριμένα κατά κύριο λόγο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να υπάρξει αλλαγή του κανονισμού. Και είναι και ζήτημα πολιτικό. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι από τους φυστάμενους κανόνες που λένε και θα το πω και δυστυχώς εντός αγωγικών ο ε, υπάρχει θέμα εμπιστευτικότητας και εγώ είμαι υπεύθυνο και υπόλογος σε ό,τι αφορά απόρριτες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχει στη διάθεση της ΙΟΛΑΦ. Και υπάρχει διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Αυτό συνιστά υποχρέωση. Και ο υπεύθυνο, σύμφωνα με τον κανονισμό, που αναλαμβάνω, και με βάση και την πολύ σαφή γνωμοδότηση του επόπτη προστασία των ευρωπαϊκών δεδομένων του 7 είναι ο Γενικό Διευθυντή τη Όλαφ. Αυτό είναι υπεύθυνο. Και αυτή η διαδικασία πλέον τηρείται και ακολουθείται. Το Σεπτέμβριο με την Εποπτική Επιτροπή αποφασίσαμε τα περί της ε, διαδικασίας αυτής ως προς τις λεπτομέρειες και επαναλαμβάνω δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα, δεν υπάρχουν καθυστερήσει και δεν υπάρχουν και παράπονα ή καταγγελίες από την Επιτροπή αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τιμερμάν, ο οποίος το είπε και το δήλωσε στη διάρκεια τη ακρόαση, δυστυχώ όμως το αποτέλεσμα της ακρόαση ε, πέρασε στον τύπο πάλι καλυπτόμενο από ένα πέπλο ομίχλη. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι εμείς στηρίσαμε του κανόνε, εξακολουθούμε να τηρούμε του κανόνε όπω οφείλουμε. Αν τώρα ε, πρέπει να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντως από πλευράς μας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, πρόβλημα με κανένα φάκελο. Δεν εμποδίστηκε πρόσβαση σε κανέναν φάκελο. Αυτά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Συνδεδεμένο με αυτό το ζήτημα είναι η πρόσβαση της ε, Επιτροπής Εποπτείας στην έκθεση και στα δεδομένα του φακέλου Νταλή. Τώρα δεν ξέρω πώς να το πω ότι εξεπλάγει ή κάτι άλλο έπαθα, αλλά τέλο πάντων όταν διάβασα πει επαύριο της ακρόασης αυτής κάποιες ε, δημοσιεύσεις, κάποια δημοσιεύματα στον τύπο που έλεγαν ότι η Επιτροπή δεν είχε πρόσβαση στον πλήρη φάκελο της υπόθεσης Ντάλι. Πραγματικά εξεπλάγει και όχι μόνο. Πρέπει να σας πω ότι υποφέραμε στην όλα από αυτό. Μας τύχησε, διότι και στις ε, θεσμικές συναντήσεις ε, εδώ με το Κοινοβούλιο επαναλήφθηκε αυτό το σχόλιο. Θέλω όμως να είμαι ε, πιστός στην πραγματικότητα και μόνο αυτό. Θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή Εποπτείας ακριβώς με βάση τις διευθετήσεις εργασίας που είχαμε συμφωνήσει μαζί τους και είχε υπογραφεί και από τη δική τους πλευρά αυτή η συμφωνία ότι σε πρώτο βαθμό παίρνουν ε, την σύντομη εκδοχή της έκθεσης χωρίς καν να χρειάζεται να τη ζητήσουν. Την παίρνουν αμέσως. Μετά όμως ζήτησαν πλήρη πρόσβαση ε, στην υπόθεση. Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα ακριβώς, 17-18 του μήνα, ακόμη και πριν δηλαδή ε, στείλουμε στη Μάλτα την υπόθεση αυτή, πήραν όλα τα στοιχεία. Όχι η Κομισιόν, για να το πω και αυτό, γιατί δεν ε, δικαιούται, δεν εξοδοτείται, η Επιτροπή Εποπτείας είχε όμως πρόσβαση άμεσα στον πλήρη φάκελο όπως είχε ζητήσει. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ήταν στα χέρια του ο φάκελος μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για 1,5 μήνα, όπως ζήτησαν. Δεν υπάρχει και κάτι περίεργο σε αυτό, γιατί το γράφει η συμφωνία μας. Αυτή ακριβώς είναι και η διαδικασία που θα έλεγα ότι επιβάλλεται μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Εποπτείας. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά εκπλήσωμαι ε, μετά την ακρόαση ήταν σαν να μην έγινε αυτό και σαν να πήραν μόνο την σύντομη εκδοχή. Λοιπόν, θέλω να τα ξεκαθαρίσω όλα αυτά τα πράγματα, διότι είναι πραγματικά στοιχεία. Και ελπίζω, ακόμη κι αν είναι κάπως αργά, να συνεισφέρω στη διάλυση αυτής της ομίχλης. Και τώρα, αν με επιτρέπετε, θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα, που επίσης ε, ετέθη ότι ο Γενικός όλα Όλαφ δηλαδή δεν τήρησε τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής Αποπτίας. Ξέρετε, εξακολουθώ να έχω δυσκολίες. Δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτό, τι εννοεί. Εγώ πρέπει να σας πω ότι του σέβομαι. Σέβομαι την Επιτροπή απόλυτα, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς εγώ δεν μπορώ να του σέβομαι. Διότι δεν επιβάλλουν καμία υποχρέωση στην Όλαφ ή στο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Άρα πώς να μην σεβαστώ κάτι που δεν υπάρχει. Να μην σεβαστώ τους κανόνες π.χ. των Γερμανών ελεγκτών. Οι εσωτερικοί διαδικαστικοί κανόνες δεν αναφέρονται στον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Μη μου αποδίδεται λοιπόν υποχρεώσεις ή ουδήποτε τύπου. Είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να καταλάβω πώς δεσέβομαι τους κανόνες ή πώς παραβιάζω τους κανόνες εφόσον δεν υπάρχει καμία υποχρέωση παρουσίας ή συμμετοχής της όλα στο συγκεκριμένο. Δεύτερον, ακόμα και αν υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις από πλευράς της Όλαφ στους κανόνες, η, ε, θα έλεγα οι, οι δυνατότητες αυτές δεν θα ήταν νομικά δεσμευτικές. Καταλαβαίνετε ότι ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ενός σώματος δεν ισχύει για τα άλλα σώματα. Εμείς έχουμε τον δικό μας κανονισμό με συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν μόνο για την όλα όχι για σας ή για οποιοδήποτε άλλο όργανο. Αυτά και έχουμε στο τελευταίο σημείο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω περισσότερο από αυτά τα οποία σας παρουσίασα μέχρι τώρα. Θέλω όμως να είμαι όσο περισσότερο γίνεται συγκεκριμένος και δεν θα ήθελα να περάσω σε ιδεολογικού τύπου ή θρησκευτικού τύπου συζητήσεις. Σέβεστε το συγκεκριμένο, ε, πιστεύετε στο συγκεκριμένο ή τα λοιπά. Όχι, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του απάντηση εκεί. Εγώ προφανώς και σέβομαι του συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αλλά νομίζω ότι η Όλαφ αντιμετωπίστηκε με πολύ αρνητικό τρόπο, γιατί τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε και αυτά τα οποία υπόθηκαν στο Κοινοβούλιο και πήγαν και στις εφημερίδες, ότι εγώ παραβιάζω κανόνες, ότι εμείς δεν σεβόμαστε στην Όλαφ κανόνες, είναι κάτι το δυσάρεστο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι σεβόμεθα ή δεν σεβόμεθα τους εσωτερικούς κανονισμούς ενός άλλου οργάνου. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω μαζί σας για να μην υπάρχουν παρανοήσεις στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, σέβομαι τους κανόνες κανόνες όμως οι οποίοι δεν είναι δεσμευτικοί για την Όλαφ. Οπότε ακόμα και αν ήθελα να παραβιάσω τους κανόνες αυτούς που δεν θέλω να το κάνω έτσι κι αλλιώς δεν είμαι σε θέση να το κάνω. Ας πούμε ότι εγώ αποφασίζω να παραβιάσω τους δικούς σας κανόνες. Ε, δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Λοιπόν, για τα θέματα προσωπικού. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο πραγματικά σημείο ίσως για μένα να μην είναι ένα τόσο τρομερό θέμα, να μην είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ίσως η Ελεγκτική Επιτροπή στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι πιο υπεύθυνη απέναντι σε τέτοιου είδους θέματα. Είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό και στο παρελθόν με το Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται. Η γραμματεία της Επιτροπής αυτής, εδώ και 13 χρόνια που λειτουργεί, ποτέ, ποτέ επαναλαμβάνω, δεν είχε το δικό της προσωπικό. Είχε τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα τρία-τέσσερα χρόνια ή πέντε χρόνια, είχε τέσσερις-πέντε δικούς της υπαλλήλους. Κάποια στιγμή έφτασαν στους επτά. Τώρα μου λένε ότι εγώ ε, έκοψα τον αριθμό αυτό, ε, έδιωξα ε, δύο ανθρώπους, δύο μέλη του προσωπικού για να μην ελέγχομαι, υποτίθεται. Αυτή ήταν η πρόθεση που μου αποδόθηκε. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ όχι επαναλαμβάνω, σέβομαι τον κανόνα λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, αλλά η ίδια η Ελεγκτική Επιτροπή, ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικός για μας. Πιστεύω στον θεσμικό ρόλο που έχει η Ελεγκτική Επιτροπή. Όχι μόνο είναι σημαντική πολιτικά, αλλά είναι απαραίτητο η Επιτροπή αυτή να προστατεύσει την ανεξαρτησία της ΟΛΑΦ και να δίνει τη δυνατότητα στην ΟΛΑΦ να είναι πραγματικά υπόλογη προς τα έξω. Το να μου λέτε ότι έδιωξα εγώ δύο ε, για να κάνω τη ζωή τους δύσκολη ή για να αποφύγω κάποιες μορφές ελέγχου, να μην υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος, ε, αυτό δεν είναι σωστό και, και, και σε επίπεδο γεγονότων αυτό το οποίο έχει συμβεί δεν είναι αληθές και σε επίπεδο προθέσεων αυτό το οποίο μου αποδίδεται είναι επίσης λάθος. Και σε σχέση με το οργανόγραμμα, εγώ απλά πήρα από το οργανόγραμμα αυτό δύο κενές θέσεις, κενές, ε, για αρκετά χρόνια κενές. Και τις χρησιμοποίησα για την ερευνητική υπηρεσία της ΟΛΑΦ. Αυτό έκανα. Δηλαδή στην ουσία εγώ αφαίρεσα τη δυνατότητα από την Ελεγκτική Επιτροπή να έχει στη διάθεσή της 8 άτομα. Δεν είχε ποτέ 8 άτομα, θεωρητικά μιλάμε. Αλλά στην ουσία πήρα δύο κενές θέσεις και τις μετέφερα στον τομέα της έρευνας. Αυτό έκανα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται η διαμεσολάβηση του Κοινοβουλίου γύρω από τα θέματα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλησα να σας εξηγήσω τι έγινε. Εγώ δεν έκοψα θέσεις εργασίας, δεν ήταν κατηλημένες αυτές οι θέσεις. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτή τη φάση έχω πάρα πολλές δυσκολίες να δώσω δύο επιπλέον θέσεις στη γραμματεία. Αναφέρθηκα και στις δύο τελευταίες συναντήσεις τις οποίες είχαμε εδώ. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση για πρώτη φορά, σαν Όλαφ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, για 13 χρόνια δηλαδή, να μειώσουμε το προσωπικό μας, όχι μόνο η Όλαφ, αλλά όλες σχεδόν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για λόγους τις οποίες γνωρίζετε σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή καλά. Οκτώ θέσεις λιγότερες, 2% στον προϋπολογισμό μας λοιπόν φέτος και 1% το οποίο θα γίνει τον επόμενο χρόνο ίσως και 2% πάλι. Οπότε ε, θα πρέπει να διώχνουμε 8 κατέτος, στην ουσία δηλαδή στα 5 χρόνια 40 άτομα. Είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό του προσωπικού κατά 23, αλλά ίσως να φτάσουμε και στο 40. Και αν τα πράγματα χειροτερεύσουν, ίσως να καταλήξουμε και σε χειρότερες καταστάσεις. Ταυτόχρονα η ΟΛΑΦ έχει φτάσει στο μέγιστο δυνατό ποσοστό αν θέλετε υποθέσεων που έρχονται προς έρευνα σε μας. 30% περισσότερες φέτος από πέρυσι που πέρυσι ήταν το ιστορικό ρεκόρ για τις υποθέσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, εμείς μειώνουμε το προσωπικό και αυξάνουμε τον κύκλο εργασιών μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι συνθήκες λειτουργίας για μας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Λοιπόν, τελειώνω με κάτι σχετικά θετικό. Μίλησα με τον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής πριν λίγες μέρες. Καταλήξαμε νομίζω σε μια κάποια συμφωνία και θα ξεκινήσουμε μια από κοινού πρωτοβουλία προς τα υπόλοιπα όργανα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα της μείωσης του προσωπικού της ΟΛΑΦ. Η μείωση του προσωπικού της ΟΛΑΦ επηρεάζει αρνητικά και τις δυνατότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής να κάνει καλά τη δουλειά της. Και ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά και τις ερευνητικές ικανότητες τις οποίες έχει η ΟΛΑΦ. Ελπίζω λοιπόν αυτές οι διευκρινήσεις να βοήθησαν όχι μόνο στο να ξεκαθαριστούν κάπως τα πράγματα, αλλά για να μπορέσετε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η ΟΛΑΦ ασχολείται με την υπόθεση αυτή. Εμείς σαν ΟΛΑΦ θέλουμε μια σωστά λειτουργούσα ελεγκτική επιτροπή. Θέλουμε να εργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να έχουμε και την δική σας αμέριστη συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Κέσλα από την πλευρά της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θέλω να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις. Ως Επιτροπή είμαστε η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες να πληροφορηθούμε για ορισμένα θέματα. Η όλα φυσικά είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και σεβόμαστε το ρόλο της ΟΛΑΦ βέβαια και την ανεξαρτησία του, αλλά σε μια δημοκρατία πρέπει ακόμα και ανεξάρτητοι φορείς να εμπλέκονται σε μια διαδικασία διασταυρούμενων ελέγχων. Γι' αυτό η... δημιουργήθηκε και η Επιτροπή Παρακολούθησης. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά το θέμα αυτό όταν ε, μέλη της ε, εποπτικής αυτής επιτροπής αναφέρουν σε δημόσιες συνεδρίασεις ότι βλέπουν να περιορίζεται η δυνατότητα δράσης τους. Γι' αυτό η Επιτροπή μας αποφάσισε να υπάρξει αυτή η δυνατότητα η Επιτροπή η Εποπτική να είναι παρούσα σε μια κοινή συνεδρίαση μαζί σας, κύριε Κέστερ. Η Επιτροπή η Εποπτικού Χαρακτήρα βέβαια δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Δεν θέλουμε αυτό να το αναβάλουμε στο διενικές, αλλά εμείς θεωρούμε ότι εξακολουθεί να είναι επιθυμητό να υπάρξει αυτή η δυνατότητα να ακούσουμε και την άποψη της Εποπτικής Επιτροπής και επομένως να εξασφαλίσουμε ότι η επιθυμία της Επιτροπής μας θα μπορέσει να υλοποιηθεί, δηλαδή να ακούσουμε και εσάς και την Εποπτική Επιτροπή. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ θα αρχίσει στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο αρχικά γιατί ήθελα να πω ότι τουλάχιστον ε, εγώ δεν έχω λάβει αυτές τις απαντήσεις του κυρίου Κέσλερ. Νομίζω τους ε, έλαβαν οι συντονιστές, όχι όμως οι υπόλοιποι βουλευτές. Ο κύριος Κέσλερ πολύ καλά μας τα εξήγησε και κατάλαβα ε, τι απαντήσει έδωσε σε τι ερωτήσεις, για ποιου λόγους. Όμω, πρόσβαση εγώ προσωπικά δεν είχα σε απαντήσεις αυτές του κυρίου Κέσλερ. οπότε θα περιοριστώ αυστηρά στις πληροφορίες που έλαβα τώρα διαστόματος του κυρίου Κέσλερ. Και βέβαια ότι ακούσαμε στην ακρόαση και στην πρώτη την κεκλεισμένη και στην άλλη. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο κύριος Κέστρα είχε κάθε συμφέρον και ε, οφείλει να μας δώσει όλε αυτές τις πληροφορίες. Τώρα ξέρω ακριβώς τι πληροφορίες έδωσε αφού δεν τις έχω, έχω λάβει, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω την ανησυχία του και θα ήθελα απλά να σας πω κύριε Κέσλερ ότι δεν μας εκπλήσει το γεγονό ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα έρχεται από την Επιτροπή Αποπτείας ε, κάποια καταγγελία, και σίγουρα ε, μας ενδιαφέρει και μας ανησυχεί. Γιατί νομίζω ότι και εσείς αρχικά είχατε εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις όταν παρουσιάσετε τα πράγματα. Τέλος πάντων, ο διευθυντής ή η διευθύντρια, αν ποτέ υπάρξει θα δούμε, της Όλαφ Σίγουρα κάποιες φορές έχουν κάποιες εντάσεις με την Επιτροπή Εποπτείας, αλλά το θέμα είναι ότι για μας αυτή η Επιτροπή Εποπτείας έναν τόσο πολύπλοκο ε, οργανισμό όπως είναι η Όλαφ, που εξακολουθεί να έχει πολλές αδυναμίες σε, σε πολλούς τομείς. Άρα η Επιτροπή Εποπτείας είναι εγγύηση αυτής της έντασης και αυτής της προσοχής που πρέπει να δείχνει για να μην έχουμε ολιστείς και εκτροπές από την πλευρά της ε, Ολαβάρα, οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, στοιχείο που μας ε, θέτει υπόψη μας η Επιτροπή Εποπτείας μας ανησυχεί και φυσικά πρέπει να το ερευνήσουμε. Θα σας ρωτήσω το εξής. Μας λέτε ότι από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο, για 7 μήνες δηλαδή, λόγω της οργάνωσης, της αναδιοργάνωσης, υπήρχαν προβλήματα. Τι προβλήματα είναι το απλό ερώτημα δεν ε, δίνατε τις εκθέσεις, τους φακέλους, γιατί από ό,τι κατάλαβα η νέα αυτή η συμφωνία ισχύει από τον Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά τι έγινε από το Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ίσχυαν ό,τι ίσχυε μέχρι πριν. Τι... Υπήρχαν καθυστερήσεις. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πήραν αυτά που ήθελαν, δεν ξέρω, τι επέστρεψα. Τι προβλήματα υπήρξαν ακριβώς αυτούς τους 7 μήνες από το Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Γιατί και αυτό μας ανησυχεί. Και φυσικά ε, θέλουμε να ξέρουμε ότι όλα έχουν πλέον διευθετηθεί, αλλά τι έγινε αυτό το εφτάμινο. Έπειτα, ξέρετε πολύ καλά ότι το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας εξαρτάται από την απόφαση του διευθυντή της Όλαφ. Έχουν ή δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό, γιατί την αρμοδιότητα τη τελέχωσης την έχετε εσεί και πριν ο προκατοχό σα. Η Επιτροπή Εποπτείας είχε 7 το πολύ άτομο προσωπικό. Τώρα τι είναι αυτή, είναι διοικητική πάλι, τι είναι ακριβώς. Και τώρα θέλω να μου πείτε, αυτοί που έχουν τώρα τι είναι ακριβώς, σε ποιο βαθμό, ε, ποιο βαθμό έχουν και αυτά τα δύο άτομα. Ήταν διοικητική πάλι τι ήταν, που, υπάλληλοι διοίκηση τι ήταν. Πέντε, π.χ. είναι υπάλληλοι διοίκηση. Ποιοι από αυτού ήταν υπάλληλοι, διοίκηση, ποια ήταν η διοίκηση κτλ. Το θέμα είναι να είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους και να κάνουν ε, την εποπτεία και να είναι και ανεξάρτητοι βέβαια. Και αποτελεσματικοί τέλος, όσο σας ρωτήσω. Μας μιλήσατε και για την ομίχλη και για τον τύπο και τα δημοσιεύματα που βγήκαν. Πρέπει να έχετε υπόψη σας στην περίπτωση του κυρίου Ντάλι, που είναι ένα θέμα που πήρε ε, πολλά φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Είναι λογικό. Εμάς μας λέτε μετά πιέσει ότι υπήρξαν. Τι πιέσει υπήρξαν. Το πρώτο, ο πρώτος που βγήκε ε, στα ΜΜΕ ήταν εσείς. Και είχαμε και αυτές τις συναντήσεις. Και εγώ έχω και κάποιες πληροφορίε από τη συνέντευξη τύπου που κάνατε εσείς. στείλατε και τις ε, πληροφορίε και το φάκελο, είπατε στις Μαλτέζικε αρχές, Τέλο πάντων, ε, είπατε όμω για πιέσει, δεν ξέρω περί τίνο πρόκειται. Και τελικά δημιουργείται ολόκληρη χιονοστιβάδα από όλα αυτά. Εσεί είστε, είπατε, υπόλογο για την εμπιστευτικότητα και για την εχεμήθεια. Όταν όμω βγαίνουν τα πράγματα στα ΜΜΕ, εντάξει, άλλο είναι η διαφάνεια, άλλο είναι να υπάρχει υπερβολική κάλυψη από τα ΜΜΕ, υπερβολική προβολή. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ελέγξουμε το τι βγαίνει προς τα έξω στον τύπο για να μην δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, αυτή η χιονοστιβάδα αν θέλετε, για θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης ε, για καλό για κακό λόγο. Πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ χρειάστηκε να δω ένα ε, ζήτημα για τον ορισμό μελών του του Τέλο πάντων, εκεί ασχολήθηκα. Δεν έχω ιδιαίτερα εντρυφήσει, αλλά τέλο πάντων. Και έχω και ένα ακόμη θέμα που θέλω να σα ε, ρωτήσω. Για την αναδιοργάνωση. Από τέσσερι ε, διευθύνσει η Όλαφ πλέον έχει πέντε και έχει και μία μονάδα συντονισμού. Κάνατε αυτή την αναδιοργάνωση λοιπόν. Το θέμα είναι πρέπει να υπάρξει νέα συγκέντρωση και εστίαση στο συντονισμό. Το να έχουμε αυτή τη μονάδα συντονισμού ουσιαστικά κάπω διασπαθίζονται οι πόροι περισσότερο, διασκορπίζονται και όχι δεν συγκεντρώνονται. Ε, τι γίνεται, δεν έχουμε ανάγκες περισσότερη έρευνα. Εκεί δεν πρέπει να σιάσετε. Σα ευχαριστώ κυρία Αγιάλα Σέντρη. Η κυρία Γκρέσλα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ Διευθύντα, εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αυτή η συνάντηση να μπορέσει να γίνει μαζί με την Εποπτική Επιτροπή. Αλλά, παρόλα αυτά, έχετε την ευκαιρία να μας πείτε τη δική σας πλευρά και θα πρέπει να ακούσουμε χωριστά από την Επιτροπή Εποπτική. Εγώ βλέπω να υπάρχουν αντιφάσεις φαινομενικά σε αυτά τα οποία λέτε. Υπάρχουν προβλήματα. Λέτε από τη μια μεριά, μετά λέτε δεν υπάρχουν προβλήματα. Είπατε ότι από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα. Και επίσης επί τη βάση αυτών που μας είπατε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η Εποπτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ένα πρώην δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ένα πρώην αστυνομικό αξιωματικό, ένα λογιστή, βουλευτέ κτλ. Ότι έχει προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα μα έχουν παρουσιαστεί και επίση έχουν δοθεί εγγράφο στα θεσμικά όργανα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι εσείς αντιτράτε μονάχα όταν είσαστε υποπίεση. Θα ήθελα να δείξετε ένα καλύτερο πνεύμα συνεργασίας. Δεν το έχετε δείξει μέχρι στιγμής εγώ. Λυπάμαι για τις δυσκολίες που υπήρξαν με την Επιτροπή Εποπτικού Χαρακτήρα έχω δει τις δυσκολίες της Εποπτικής Επιτροπής να καταλήξει σε κάποια συμφωνία μαζί σας. Τελικά αυτό δεν κατέβησε δυνατό. Σας παρακάλεσα, σας προσωπικά παρακάλεσα και τον κύριο Επίτροπο Σεμέτα. Αλλά γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει οξυνθεί τόσο η κατάσταση. Θα ήθελα πραγματικά να έχω ένα, μια απάντηση για το θέμα αυτό και σας παρακαλώ αυτή η απάντηση να είναι ελεύθερη από εσωτερικές αντιφάσεις. Είπατε επίση ότι ήρθατε εδώ από σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γιατί θέλετε να λογοδοτήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είδα τις ε, απαντήσεις, τις ερωτήσεις μας σε σχέση με την υπόθεση Ντάλι. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει σεβασμός προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εσείς πήρατε θέση ενώπιον της, ε, των μέσων ενημέρωσης και Προτού γίνει αυτό το πράγμα εναντί του Κοινοβουλίου. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι λαθασμένο. Και πρέπει να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα, γιατί ότι αυτά τα οποία είπατε περισσότερο συγκάλυπταν παρά αποκάλυπταν την κατάσταση και δεν ανταποκρινόταν στην ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πληροφορηθεί. Γιατί τι είναι η Όλαφ, είναι μια υπηρεσία που κάνει διοικητικές έρευνες. Στην περίπτωση Ντάλι έχει κλείσει αυτή η διαδικασία και τελικά οδήγησε αυτή η διαδικασία στην παρέτηση του κυρίου Επιτρόπου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο εσείς πρέπει να, δεν, ε, ε, πρέπει να αρνείστε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες. Και εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που υπάρχει με την Εποπτική Επιτροπή δεν βοηθάει καθόλου η Επιτροπή Εποπτικού Χαρά, η Εποπτική Επιτροπή θα πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά. Κανείς δεν θέλει να τον ελέγχουν, αλλά το πρόβλημα αυτό μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ και της Εποπτικής Επιτροπής το παρακολουθώ εδώ και 8 χρόνια. Πράγματι πάντα ήταν δύσκολα τα πράγματα γιατί η σύλληψη αυτής της δομής ήταν πράγματι ένα πρόβλημα. Αλλά βλέποντας πίσω αυτά τα 8 χρόνια Ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα τα προβλήματα και τόσο οξέα όσο σήμερα. Και νομίζω ότι εσείς με αυτή την όξυνση των πραγμάτων ουσιαστικά θέτετε σε δυσκολία τη δική σας θέση ως Διευθυντού της ΟΛΑΦ αλλά και την Εποπτική Επιτροπή. Είναι ένας φορέας που έχει διοριστεί από μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτός ο φορέας θα πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσετε με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή την εποπτική επιτροπή. Θέλουμε μια όλαφη η οποία είναι αποφασιστική και η οποία θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Σα παρακαλώ όμω να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και η Υποπτική Επιτροπή και θα πρέπει να συνεργαστείτε μαζί τη. Ο κύριο Γκάιερ. Δεν έχω ένα ερώτημα να σα θέσω, έχω όμω ένα σχόλιο κύριε Γενική Διευθυντά. και αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Επιτροπή μας. Εγώ θέλω να διαχωρίσετε δύο θέματα. Το ένα από αυτά είναι το ερώτημα της σχέσης μεταξύ του, του κυρίου Κέσλε και της Εποπτικής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη διοικητική αρμοδιότητα. Αυτό είναι σαφές. Εγώ χαίρομαι που μπορούμε να σας ακούσουμε χωριστά από την Εποπτική Επιτροπή γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν πολύ περισσότερα τα πράγματα και να παίξουμε το ρόλο των δικαστών όταν οι δύο πλευρές θα παρουσιάζαν τις απόψεις του. Αυτό δεν νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πολύ να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο. Η επίλυση αυτή τη τεχνικού χαρακτήρα αντιπαράθεσης μεταξύ του Γενικού Διευθυντού και της Εποπτικής Επιτροπής θα πρέπει να διαχωριστεί πλήρως από το περιεχόμενο της υπόθεσης Νταλή. Και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά τα οποία έχουν γίνει σαφή εδώ και ένα μήνα. Έχουμε συζητήσει ήδη δύο-τρεις ώρες με το Γενικό Διευθυντή στην, ε, σε στο Στρασβούργο. Υπάρχει αυτή η έκθεση και υπάρχουν δύο πηγές από τις οποίες έχει συνταχθεί αυτή η έκθεση από την Κομισιόν και από τις αρχές της Μάλτας. Έχει πάρει στοιχεία. Μπορεί εσύ να έχεις την έκθεση, εγώ δεν την έχω, λέει στην κυρία Γκρέσλε ο κύριος Γκάιερ. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα του ποιος έχει αυτή τη, την ε, έκθεση. Ζητήσαμε από την Κομισιόν να πάρουμε αυτή την έκθεση. Μας είπε η Κομισιόν όχι δεν μπορείτε να την έχετε αυτή την έκθεση. Και περιμένουμε από τον κύριο Κέσλε να μας πληροφορήσει. Αλλά πόσο καιρό λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε για να πάρουμε αυτά τα στοιχεία. Και το επόμενο ερώτημα είναι, έχουμε εμεί το χαρακτήρα μια επιτροπή η οποία είναι ερευνητικού χαρακτήρα ή όχι. Δεν είμαστε ερευνητική επιτροπή. Αλλά πρέπει εμεί να είμαστε. Εμεί είμαστε, έχουμε την υποχρέωση να παρακολουθούμε θέματα ε, στον προπολογισμό. Εμεί συμφωνήσαμε μεταξύ των συντονιστών ότι πρέπει να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει τα θέματα αυτά να τα αφήσουμε σε μια επιτροπή έρευνα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια επιτροπή η οποία έχει εντολή να ερευνήσει για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, δεν θέλω να μας αντιμετωπίσετε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι έχετε την υποχρέωση να μας παράσχετε τα απαραίτητα στοιχεία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, λέει ο πρόεδρος. Το γεγονός παραμένει. Ότι η Επιτροπή μας και αυτό παραμένει η σωστή διαδικασία να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Στις 15 Οκτωβρίου είχαμε πάρει τις πληροφορίες αυτές που δόθηκαν από εσά κύριε Γκέσλερ στην Κομισιόν. Στις επόμενη μέρα εγώ μίλησα στον Επίτροπο Σέμετα και θέλησα να πληροφορηθώ για το τι έγινε με τον Επίτροπο Ντάλι και την ίδια μέρα υπήρξε μια ανακοίνωση τύπου της Κομισιόν και στις 17 Οκτωβρίου νομίζω ότι έλαβε χώρα μια συνέντευξη τύπου της Επιτροπής όπου ήσασταν και εσείς ο κύριε Κέσλερ και μετά τα μέλη της Επιτροπής μας μετά από τη θέση που λάβατε εσείς στην Επιτροπή στην διάσκεψη τύπου έλαβαν την εντύπωση ότι ο Γενικός Διευθυντής Τη Όλαφ προτιμά να πληροφορήσει τον, τα μέσα ενημέρωσης ενώ δεν θεωρεί ότι θα έπρεπε προηγουμένως να πληροφορήσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εμείς ζητήσαμε να, ε, να, κάνει μια, να γίνει μια κοινή ε, συνεδρίαση μαζί σας και κλεισμένο των θυρών και θεωρήσαμε ότι υπήρξε μια πολιτική απόφαση από την Κομισιόν σε σχέση με την αποχώρηση του κυρίου Νταλή και γι' αυτό εμείς ζητήσαμε μέσω της συνέλευσης των Προέδρων να υπάρξει καταρχήν μια επαρκής πρόσβαση στην ε, έκθεση του, της ΟΛΑΦ τα θέματα αυτά και επίσης να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο της ε, Κομισιόν, της Επιτροπής, να έλθει ενώπιον της ε, Συνέλευσης των Προέδρων και να απαντήσει ερωτήματα. Εγώ δεν είμαι απλώ πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. είμαι και μέλος μιας πολιτικής ομάδας εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινοβούλιο στον κόσμο που μπορεί να υπάρξει <clears throat> όπου ένας υπουργό παρετείται <clears throat> χωρίς ο πρόεδρος, ο επικεφαλής αυτής της κυβέρνηση σε μια δημόσια συνεδρίαση πληροφορεί το κοινοβούλιο αυτό γιατί <clears throat> έγινε αυτή η παρέτηση του Υπουργού του. Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι διαφορετικό. Θυμάστε αυτά που είπε χθε ο πρώην καγκελάριο Χέλμουτ Σμιτ σε μια σε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και είπε ότι περιμένει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια επανάσταση στην Ευρώπη και να πάρει στα χέρια του τα ενία της... του δημοκρατικού ελέγχου. Και επομένως εμείς θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να θέσουμε το ερώτημα τι έγινε στην περίπτωση αυτή του κυρίου Ντάλι. Και αυτό είναι κάτι που θέτουμε όχι μόνο εμείς ως ερώτημα, αλλά και από την κοινή γνώμη. Όταν λοιπόν αυτό το ερώτημα δεν την χάνει απάντηση, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και δεύτερον, αν εμείς σαν άμεσα εκλεγμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν μπορεί η Κομισιόν ή η Όλαφ να μας πληροφορήσει και να μας δώσει πρόσφαση στην πληροφορία, τότε δεν είναι μοναχά το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό σαφές στην κοινή γνώμη. Έχουμε το καθήκον να πούμε στην κοινή γνώμη ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν και η ΟΛΑΦ δεν μας δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία και αυτό διότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάθε δικαίωμα οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι τους να ελέγχουν την Κομισιόν και ο έλεγχος χωρίς πληροφόρηση δεν είναι εφικτός. Αυτά λοιπόν για τη δράση της Επιτροπής μας. Υπάρχουν ε, οικοτολογίες στις οποίες εγώ δεν θέλω να συμμετάσχω. Θέλω να πάρω... Θέλω να έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορεί κάποιοι άλλοι να θέλουν να παίξουν με τις φήμες αλλά χωρίς να θέλω να αποκαλύψω πράγματα που είπε ο κύριος Μπαρόσο σε μια κλειστή συνεδρίαση, εγώ θέλω και πάλι να τονίσω ότι είπα στον κύριο Μπαρόσο ότι το καλύτερο, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι θεωρίες συνωμοσία που κυκλοφορούν εδώ είναι πράγματι η Κομισιόν η ίδια να κάνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και να εξασφαλίσει την απαραίτητη διαφάνεια. Και επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής διευκρίνηση για τη διαδικασία αυτή και να συνδέεται με μια δημόσια πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Αυτό αφορά την περίπτωση Ντάλι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ε, επίσκεψη του κυρίου Ντάλι, αλλά με αυτά τα οποία ελέγχθησαν από την Εποπτική Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου και θα θέλαμε ο κύριος Ντάλι, ο κύριος, ο κύριος Κέσλερ, να δώσει μια απάντηση και στα θέματα αυτά. Αλλά <clears throat> νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά. Συζητήσαμε με τους συντονιστές και ό,τι κάναμε το έχουμε κάνει μαζί με τους συντονιστές. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω κάνει εγώ προσωπικά ήταν να δώσω συνέχεια στην ε, θέληση του κυρίου Κέσσερ να λάβει το λόγο σε μια δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αυτό ήταν στο πνεύμα συνεργασίας. Και σας παρακάλεσα για αυτό το λόγο να απαντήσετε στα ερωτήματα των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος να δώσω κάποιες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα για την υπόθεση Ντάλι, όπως είδατε και σε αυτή τη συνεδρίαση, ήμουν πολύ πιο ταπεινόφρον από ότι εσείς. Δηλαδή, εγώ ήθελα να διευκρινίσω απλά κάτι, ότι στην περικειμένη περίπτωση όλα φτύρισε κυριολεκτικά όλους τους κανόνες και ιδίως ό,τι αφορά την Επιτροπή Εποπτείας αν ε, υπάρχει παρανόηση πάνω σε αυτό, εντάξει δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά εδώ ήρθα για να το ξεκαθαρίσω. Ότι εμείς ακολουθήσαμε τους κανόνες και τηρήσαμε τη συμφωνία με την Επιτροπή Εποπτείας. Δεν θέλω λοιπόν, δυστυχώς έγινε βέβαια, ότι συνήθισαν συμπεράσματα. Δεν θέλω να συμβαίνει αυτό όμως από το ε, απ' έξω θα καταλήγουν κάποιες ε, συμπεράσματα ότι δηλαδή Όλαφ έχει να κρύψει κάτι για την υπόθεση Ντάλι από την Επιτροπή Εποπτεία. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο και αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. I mean, Μιλάω για την Επιτροπή Εποπτεία, ναι. Δυστυχώ το σχόλιο τη κυρία Κρέσλι είναι εκτό μικροφώνου. Ναι, θα επανέλθω σε αυτό, αλλά εγώ τώρα ήρθα για να σα μιλήσω για αυτό το θέμα. Είχαμε τα αποτέλεσμα τη ακρόαση πριν από ένα μήνα και κάτι πια πράγματα που είπε η Επιτροπή Εποπτεία οδήγησαν και τον τύπο αλλά και κάποια μέλη τη Επιτροπή σα να πούν να ισχυριστούν κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή εμεί αποκρύψαμε πληροφορίε ή δεν δώσαμε πρόσβαση στην Επιτροπή Αποπτία. Ελπίζω τέλο πάντων αυτό πλέον να είναι σαφέ, έστω και ένα μήνα μετά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εγώ δεν ήθελα να τροφοδοτήσω τον τύπο απαντώντας για να έχουμε απαντήσει και ξανά απαντήσεις και συνέχεια νέα δημοσιεύματα. Προτίμησα να έρθω ενώπιον ημών της Επιτροπής σας για να σας τα εξηγήσω και να δώσω τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Εκτός μικροφώνου σχολή τη Σαγιάλα. Ναι, ναι, ναι. Για την υπόθεση Ντάλι μιλάω. Τώρα για το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο. Όχι, δεν ήταν υπόθεση Ντάλι τότε. Τι έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι βέβαια. Ναι, να σας απαντήσω και σε εσά, αλλά εν μέρει να απαντήσω και στο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε. Τι έγινε μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου. Το είπα και το ξαναλέω, έτσι πιο αναλυτικά. Πρώτον, δυστυχώς η Όλαφ δεν είχε ποτέ κάποια διαδικασία ή διευθέτηση εργασίας με την Επιτροπή Εποπτείας. Πριν αναλάβω καθήκοντα, ο προκάτοχός μου τέλο πάντων, είχε κάποιες διαδικασίες που δεν είχαν εφαρμοστεί. Άρα δεν υπήρχε διαδικασία. Δεν βοηθά αυτό. Πάω εγώ, είμαι δικηγόρο, αλλά δεν είμαι κολλημένο ε, με τη διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά, οι διαδικασίε βοηθάνε. Πώ να το κάνουμε. Είχαμε λοιπόν μετά ταυτόχρονα ε, από την 1η Φεβρουαρίου τη νέα Επιτροπή Εποπτείας και την αναδιοργάνωση της ε, δικής μας υπηρεσίας. Έχουμε λοιπόν την Επιτροπή Εποπτείας πέντε ανθρώπους που έρχονται ε, απ' έξω, που δεν έχουν ιδέα για τη διαδικασία αυτή και που κατά την άποψη μου χρειάζονται λίγο χρόνο για να βάλουν σε τάξη το μυαλό τους και να δουν τι ρόλο έχουν και πώς θα τον εφαρμόσουν. Και αυτοί ήταν λοιπόν ε, καινούργοι και εμείς είμαστε καινούργοι. Και ταυτόχρονα δεν υπήρχε και καμία διαδικασία. Και για να απαντήσω έτσι εν μέρη και στο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε, νέα προβλήματα λέει κυρία Γκρέσλε γιατί. Μα ακούστε, εσείς λέτε ότι πάντοτε υπήρχαν θέματα και κατά το παρελθόν με την Επιτροπή και τώρα έχουμε νέα προβλήματα. Και αν κατάλαβα καλά αυτό, ε, πάνω σε αυτό με ρωτάτε. Νέα και, και, και χειρότερα προβλήματα, λέτε. Μάλιστα. Ακούστε ένα μέρος της εξήγησης, προσθέτοντας αυτά που είπα, είναι ότι Όλαφ έλαβε νέες ε, αιτήσει, νέα αιτήματα από την Επιτροπή Εποπτείας που δεν είχε λάβει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, να έχει άμεση πρόσβαση στους φακέλους. Δεν είχαμε κατά το παρελθόν κάτι τέτοιο ως Όλαφ, δεν το είχαμε αντιμετωπίσει με τις έρευνες. Συγγνώμη, δεν μπορούμε, λέει ο πρόεδρο, να ε, ακούσουμε τι παρεμβάσει σα. Δεν μπορούμε να μεταφράσουμε. Λοιπόν, άμεση πρόσβαση των ε, φακέλων, στου φακέλου για έρευνε που είναι σε εξέλιξη είναι κάτι που δεν είχε ζητηθεί ποτέ πριν από την Επιτροπή Εποπτεία. Όταν λοιπόν πήραμε αυτά τα αιτήματα, έπρεπε και εμεί να ε, διαμορφώσουμε κάποια άποψη. Και γι' αυτό επί μήνε είχαμε ανταλλαγή αλληλογραφία με την Επιτροπή Εποπτεία για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και καταλήξαμε πράγματι, αλλά το Σεπτέμβριο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συμφωνία και θέλω και να ευχαριστήσω τον κύριο Τίμερμαν και όλη την Επιτροπή Εποπτείας που συνεργαστήκαμε και βρήκαμε ένα διακανονισμό που πλέον είναι κοινή συμφωνία. Από εκεί και πέρα, παραλαμβάνω, δεν, ε, δεν αντιμετωπίσαμε άλλα προβλήματα γιατί και οι δύο πλευρέ τηρούμε την συμφωνία που έχει τρία βήματα, τρία στάδια. Και είναι μια διαδικασία που, επαναλαμβάνω, μα επιβλήθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Άρα ζητάνε και τους δίνουμε πρόσβαση. Και αυτό έχει γίνει χωρίς κανένα πρόβλημα από τον Σεπτέμβριο και μετά. Πριν το Σεπτέμβριο, με νέα υπηρεσία, χωρίς να έχουν προηγηθεί τέτοια αιτήματα και εμείς να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη νομική κατάσταση, γιατί είμαστε υπόλογοι και εγώ θέλω να είμαι και είμαι υπόλογο και πιστεύω πάρα πολύ στην ευθύνη, στην λογοδοσία και σε όλα αυτά τα μέτρα. Επιτροπή Αποπτείας ε, και τα λοιπά και δημόσια κοινωνικά κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν τα μέσα που εξασφαλίζουν την λογοδοσία με δεσμεύουν, αλλά με δεσμεύουν και οι κανόνες και οι επιταγές των ελεκτικών φορέων όπως είναι ο επόπτης ε, προσωπικό δεδομένο. Τώρα. They work. They got... Τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ό,τι ζητήσει η Επιτροπή Εποπτεία το παίρνει. Ε, γιατί έχουμε αυτή τη συμφωνία πλέον, την οποία τηρούμε. Και έχουμε και μια διαδικασία που είναι πλήρω ευθυγραμμισμένη με τον κανονισμό περί προστασία δεδομένων. Και επίση πλήρω ευθυγραμμισμένη με τη γνωμοδότηση του επόπτη δεδομένων για την Εποπτική Επιτροπή του, της Όλαφ, ε, την γνωμοδότηση του 2007. Και δυστυχώ πριν το Σεπτέμβριο δεν τα είχαμε αυτά, τώρα όμω τα έχουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω. Και για την κυρία Σέντερ. Ίσως κατάλαβα τις απαντήσεις, αλλά παρόλα αυτά ζητάτε ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από μένα και εγώ δίνω την απάντηση στην Επιτροπή και η Επιτροπή ε, προωθεί τις απαντήσεις σε εσά που θέσατε τα ερωτήματα. Και εμεί θέλουμε να είμαστε υπόλογοι. Είμαστε υπόλογοι. Και παρόλα αυτά δεσμευόμεθα από συγκεκριμένους κανόνες και από τον νόμο. Δεν μπορώ εγώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεσμεύομαι λοιπόν και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις γιατί αφορούν την ουσία της έρευνας και δεν έχω την δυνατότητα να σας δώσω ερωτήσεις. Θέλω να διαλύσω τις παρανοήσεις και ό,τι δυσνόητο. Εγώ δεν έλαβα οδηγίες από κανέναν όπως είπαν ορισμένοι και δεν πιέστηκα από κανέναν. Δεν ένιωσα να πιέζομαι από κανένα. Δεν αναφέρθηκα σε πιέσεις προς τον τύπο. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε πιέσεις που μου ασκήθηκαν στη διάσκεψη τύπου. Και αν αναφέρομαι σε πιέσεις, αναφέρομαι στην πίεση της κατάστασης που με υποχρεώνει μετά το κλείσιμο της έρευνας, μετά την παρέτηση του Επιτρόπου, οδηγήθηκα να στείλω την έκθεση της δικαστικής υπηρεσίας της Μάλτας, να ζητήσω μάλλον αυτήν την έκθεση ε, με κατεπήγοντα τρόπο. Νομίζω ότι αυτό ήταν απαραίτητο και έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, συνάδελφοι... Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ κύριε Κέσσελ. Έχει τελειώσει η διερμηνία. Πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχω δύο συναδέλφους στον κατάλογο, την κυρία Αντρέσεν και τον κύριο Γκάιερ. Συνεχίζουμε για πέντε λεπτά στα αγγλικά λοιπόν.